meine Damen und Herren. Κυρίε και κύριοι, σα καλωσορίζω και τον κύριο Σαλαφράγκα. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα σα. Ε, έχουμε κοινή συζήτηση στο σημείο 9 και 10. Καταρχάς, θα μας παρουσιαστεί η μελέτη σχετικά με την πρόθεση μιας ευρύτερης διακρατικής ιστορικής σχέσης. Θα πάρει το λόγο ο εμπειρογνώμονάς μας. Ο καθηγητής Eric Jones και η μελέτη εστιάζεται κυρίως στους τομείς ε, στενότερης ε, συνεργασίας διατλαντικής συνεργασία και εντοπίζει σχετικού μηχανισμούς προώθησης της συνεργασίας Αυτή Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δώσουμε μια νέα διάσταση στη συζήτηση αυτή μετά την ομιλία του Ομπάμα και τις σχετικέ αντιδράσεις που προέκυψαν από πλευρά της Ευρώπης. Και παράλληλα, ο συνάδελφο Μίλαν θα μας ε, παρουσιάσει για το ίδιο θέμα, τη δική του τοποθέτηση. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά από κοινού. Να δώσουμε το λόγο καταρχάς προτείνω στον καθηγητή Jones και μετά να κάνει μια εισαγωγή ο συνάδελφος Μίλαν Μον για να συζητήσουμε από κοινού τα θέματα αυτά. Για να αποφύγουμε τις ε, διπλές δηλώσεις. Κυρία Jones, καθηγητά Jones, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ είχα μια μεγάλη συζήτηση με την Βάντα ε, σήμερα το πρωί, γιατί ανησυχούσα ότι οι διερμηνείς δεν θα καταλάβαιναν τα τεξανικά μου. Έγραψα λοιπόν την ομιλία μου. Ξέρω ότι αυτό θα κάνει την παρουσίαση λιγότερο ενδιαφέρουσα, αλλά θα κάνει τη δουλειά του των συναδέλφων σαν πιο εύκολη. Καλημέρα σας λοιπόν και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω προ την Επιτροπή σας. Είναι τεράστια τιμή το ότι μιλώ μπροστά στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρώ να σας πω μάλλον ότι η παρουσίαση αποτελεί μια κοινή προσπάθεια με συμβολή ε, διαφόρων ιδρυμάτων και εμπειρογνωμόνων ε, και στην ε, Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στη Λατινική Αμερική και επίσης να πω ότι έχω χρησιμοποιήσει και την Επιτροπή ΑΦΕΤ και τη Σουάντα και τον Τελφίν και του εισηγητή για το θέμα αυτό και χαίρομαι που έδωσαν τόσο μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό. Τι θέλω να κάνω στο χρόνο που έχω στην διάθεσή μου, να σα δώσω μια επισκόπηση τη ε, παρουσίας και των πορισμάτων τη ε, Το πλαίσιο δεν θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επίκαιρο. Στι 12 Φεβρουαρίου, στο State of the Union, στην ομιλία του, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρο τη Αμερική, ανακοίνωσε την ε, φιλοδοξία του να προωθήσει μια ευρύτερη διεθνική σχέση και εταιρική σχέση. Και την επόμενη ε, ημέρα συνήλθε με τον Χερμάν Φαν Ρόμπαϊ και τον ε, κύριο Μπαρόσο, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, για να συζητήσουν ενδεχόμενη εμβάθυνση της διεθνικής σχέσεις. Βγαίνει ο στόχος αυτός και ελπίζω να υπάρχει η πολιτική βούληση για να σημειωθεί σημαντική πρόοδο στην υπόλοιπη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Κάρλ Τεχούχτ, επίτροπος για το εμπόριο και ο ομόλογός του από πλευρά ε, Αμερικής, κ. Κόρκα, έχουν στενές σχέσεις και έχουν ε, επιδείξει τι μπορούν να πετύχουν με κοινή ηγεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα σε ό,τι αφορά θέματα ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να επωφεληθούμε από την αποφασιστικότητά τους και να αναπτύξουμε το έργο τους. Και στα πιο αισιόδοξα σενάρια παρόλα αυτά, η στενότερη σχέση με τις χώρες της Βόρειας Αμερικής δεν θα αρκέσει για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Θα αποτελέσει στην καλύτερη περίπτωση μία βάση και σε ό,τι αφορά την ε, διατλατική εταιρική σχέση και σε ό,τι αφορά την έμφαση που δίνεται στις επενδύσεις και στο εμπόριο. Η πραγματική πρόοδος θα προαπαιτήσει ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη παγκόσμια οικονομία για συνεκτική ε, ασφάλεια προς τη δημοκρατία, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερους φορείς. Θα πρέπει να σκεφτούμε και ποιες είναι οι παράπλευρες συνέπειες της παγκοσμίας παγκοσμιοποίησης, η οικονομική ενσωμάτωση υπόσχεται πολλά σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργεί και συνθήκες ε, αποστοφεροποιητικές για τις ε, πολιτικές, τα πολιτικά ιδρύματα και που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε πέρα από την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Πέντε θέματα έχει η παρουσίασή μου. Καταρχάς καταγράφουμε τι γίνεται στι ατλαντικές σχέσει και τη σχέση εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ΗΠΑ. Ε, και στο δεύτερο τμήμα ε, θα σας παρουσιάσω πιο πολύ ε, τις σχέσεις μεταξύ των νοτίων ε, χωρών Αφρικής, Κίνας και το καθεξής. Ε, στο τρίτο τμήμα μιλάω για τη σύγκληση της πολιτικής σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και βιωσιμότητας μεταξύ των χωρών ε, συνεργασία συνεργασίας. Στο τέταρτο θέμα παρουσιάζω άλλα θέματα και στο πέμπτο θέμα καταλήγω σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις. Στο αρχικό σημείο. Είναι γνωστό και επαναλαμβάνεται από την ομάδα υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ΕΕΠΑ για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό της ε, output της, ε, της παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η σχέση μεταβάλλεται ταχύτατα. Πριν από μία δεκαετία μόλις ήταν πολύ μεγαλύτερη αυτή η εταιρική σχέση. Ωστόσο αυτή η μεταμόρφωση δεν είναι πανομοιότυπα σε όλους τους τομείς. Διαφέρει ας πούμε στην ε, παραγωγή από τη, στην παροχή υπηρεσίας και επίσης ε, από το εμπόριο στις επενδύσεις. Ωστόσο το σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι Ακόμα και μια τέτοια βαθιά οικονομική σχέση ε, υπόκειται σε μεταβολές και παραδόξως η σχέση μεταξύ Βορρά και Νότου, μεταξύ ε, ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού φαίνεται ότι είναι πιο ανθεκτική και αυτό εν μέρη ίσως να οφείλεται στην παράδοση της απεικιοκρατίας και ίσως και στις εξαρτήσεις που διατηρούνται μέσω των Γενικών Συστήμα προτιμόμενων ε, ε, εμπορικών συναλλαγών. Οι χώρες της Αφρικής έχουν την τάση να ασκούν εμπορίο με την ε, Ευρώπη και υπάρχει και ιστορική διάσταση με, τις, με τους Πορτογάλους για παράδειγμα που έχουν σχέση με την Βραζιλία, με τους Ολλανδούς, τους Βρετανούς, τους Γάλλους που έχουν σχέση με την Καραϊβική. Φυσικά όλα αυτά δεν είναι απόλυτα χρειάζεται και ένα πλαίσιο για την ε, συντήρηση αυτού του προτιμόμενων εμπορικών συνθήκων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιστορικές ε, χώρες ε, με τις ιστορικές μας στην Καραϊβική, στην Αφρική και στην Καραϊβική. Η συνθήκη του Κοτονού βασίζεται στην, στις εξαιρέσεις που παρήλθαν το 2007 η οικονομική συνεργασία και οι σχετικές συμφωνίες είναι σημαντικές και χρειάζεται να κοιτάξουμε τις ε, απαιτήσει και τις ε, ανάγκες των ε, λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Αυτές οι συνθήκες και αυτές οι διευθετήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, γιατί όλες αυτές οι εξαιρέσεις έχουν ε, τύχη κατάχρηση και σε μονομερές και σε πολυμερές επίπεδο. Και τώρα συζητάμε να περάσουμε πέρα από το κοτονού πριν ε, παρέλθει το 2020 και συζητάμε να αφήσουμε την ε, ορισμό των χωρών ΑΚΕ και να βρούμε έναν ορισμό που να ταιριάζει πιο πολύ με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην εξαρτάται τόσο από την αποκεκρατική ιστορία των χωρών αυτών και μια νέα σχέση μεταξύ των χωρών του Νότου, μεταξύ των αναδυόμενων χωρών της Λατινικής Αμερικής, στην Ασία και στην Αφρική, έχει, ε, έχει λάβει πολύ μεγαλύτερη διάσταση. Και εδώ περνάμε στο δεύτερο τμήμα της ομιλίας. Σε σχέση με την διείσδυση των αφρικανικών αγορών και των ασιατικών, στην Ασία, στις αναδυόμενες δηλαδή χώρες. Μέχρι το 2009 φτάνουμε σε ένα 20% του ογκού συναλλαγών. Όσο αφορά την ε, ε, Κίνα, Βραζιλία, ε, Ινδία, Τουρκία, δεν βρίσκονται πολύ πίσω. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην Ινδία περισσότερο, που είναι μια αναδυόμενη αγορά. Η Ινδία αφορά το, έχει διεισδύσει στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αφρικής ιδιαίτερα και σύμφωνα με μία πρόσφατη δημοσίευση θεωρούμε ότι ο Νότιος Ατλαντικός θα βρίσκεται στην εμβέλεια, σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια ως προς την ε, διείσδυση της Ινδίας. Και αυτό αφορά και τις ε, πρώην απικίες της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βρεθούν ε, σοβαροί σύμμαχοι για να αντιμετωπίσουμε τον ε, κίνδυνο αυτής της νέας διείσδυσης και της ε, Κίνας. Θα πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε την παραδοσιακή εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και ΗΠΑ για να συμπεριλάβουμε και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έτσι θα ήταν δύσκολο, έτσι θα ήταν ευκολότερο με συγχωρείτε, να αντιμετωπίσουμε την Κίνα και άλλες αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Ινδία. Όμως, μία ευρύτερη διατλαντική σχέση δεν θα πρέπει να είναι καθαρά αμυντικής υφής. Θα πρέπει να συμμετέχουν οι πάντες. Και εδώ φτάνω στο τρίτο τμήμα της παρέμβασής μου, όπου θα ήθελα να τονίσω μία τάση σύγκλησης τάσης μεταξύ Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής και Λατινικής Αμερικής. Καταρχήν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια η πειρατεία στον κόλπο της ε, Γουινέας, τα συμβατικά όπλα που υπήρχαν στη Λιβύη και χρησιμοποιούνται και τα όπλα μαζικής καταστροφής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις απειλές αυτές. Η πειρατεία στον κόλπο της Γουινέας έχει αυξηθεί απειλητικά και απειλεί πολλούς παραγωγούς της Δυτικής Αφρικής. Αυτή η πειρατεία ανθίζει ακριβώς επειδή υπάρχει αστάθεια και αδυναμία. Και αυτό οφείλεται στις εμπόλεμες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες τώρα έχουν πρόσβαση σε πολλά ε, όπλα και οπλικά συστήματα. Η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής είναι επίσης μία σοβαρή απειλή και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση του θέματος. Μιλάμε για το πρόγραμμα που ε, προωθείται στον κόλπο της Γουινέας πρωτίστως και θα πρέπει να ενισχύσουμε και την παγκόσμια διάσταση μη διάδοσης όπλων μαζικής ε, καταστροφής ως προς την ενέργεια και το περιβάλλον θα πρέπει να δούμε τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και το Μεξικό που είναι βασική παραγωγή και τη Βραζιλία και τη ΣΥΠΑ που είναι ενδυνάμει παραγωγή. Έτσι μπορούμε να προωθήσουμε το εμπόριο διατλαντικά, κάτι το οποίο θα είναι ευεργετικό για όλους και μπορεί να ε, εξασφαλίσει και την ε, ασφάλεια των ενεργειακών πηγών, την ενεργειακή εξασφάλιση δηλαδή, για να έχουμε εύρωστα δίκτυα ε, ως προς τη χρήση του φυσικού αερίου. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της εξόριξης μεταφοράς και επεξεργασίας δίλησης. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο ενθουσιώδης όλοι οι εταίροι. Θα πρέπει όμως να υπάρξει σωστός επιμερισμός των δαπανών για τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για δαπάνες οι οποίες ε, πέφτουν στις πλάτες της χώρες του Νότιου Ατλαντικού. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση και εδώ φαίνονται και τα σημάδια της, ε, το αποτύπωμα μάλλον της ε, παγκοσμιοποίησης. Το οργανωμένο έγκλημα είναι ευρέως γνωστό, ιδιαίτερα σε σχέση με την ε, διάδοση και μεταφορά ναρκωτικών. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μία ολίσθηση αυτών των τάσεων. Στις ΙΠΑ, η ΙΠΑ καταναλώνουν τέσσερις φορές περισσότερο κοκαίνη από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι αντιστρέφεται αυτή η τάση. Το ίδιο αφορά και τη Λατινική Αμερική, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει και κατάχρηση και χρήση και ευρεία χρήση ναρκωτικών και αυτό αφορά και την Αφρική και την ε, Καραϊβική που αποτελούν ε, σημεία διασύνδεσης για το, την διάδοση των ναρκωτικών και το ξέπλυμα χρήματος. Πολύ, ε, πολύ, πολύ μεγάλο μέρος της δραστηριότητας προωθείται σε αυτές τις περιοχές και αυτό αφορά ιδιαίτερα το, το εμπόριο γυναικών ή δουλεμπόριο που προέρχεται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την παράνομη μετανάστευση σε διατλαντική εμβέλεια και θα πρέπει να βρεθούν συνέργειες προς αυτό. Μιλάμε για προαπαιτούμενα και προαπαιτήσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει η καλύτερη ροή πληροφοριών πρωτίστως. Και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που οθούν τους εργαζόμενους να μεταναστεύουν παράνομα για να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτή η ενδυνάμη σύγκληση πολιτικής ε, έχει μία, ενέχει μία συνέργεια και αλληλοσύνδεση και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημεία τομής. Θα πρέπει να προωθήσουμε συλλογική δράση για να προωθήσουμε τις διατλαντικές ε, σχέσεις σε φόρα διάδρασης ε, διατλαντικός. Και εδώ φτάνω στο τέταρτο τμήμα της ομιλίας μου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το δυναμικό που υπάρχει ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική. Και αυτό για δύο λόγους. Η Λατινική Αμερική δεν έχει μία επικεφαλής χώρα. Η Βραζιλία είναι η πρώτη σε πληθυσμό, έχει πολλούς πόρους και διπλωματικές αρμοδιότητες και είναι ένα σημαντικός εταίρος και για την Ευρώπη και για τις χώρες της Βορείου Αφρικής. Δεν θεωρείται όμως ότι έχει αρχηγική θέση, παρόλο που εγκρίνουμε, καταλαβαίνουμε τα προσόντα που διαθέτει αυτή η χώρα θα πρέπει ε, να δούμε κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μία ενιαία φωνή για τη Λατινική Αμερική. Η περιφερειακή ε, ηγετική θέση, θα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνονται περιφερειακές ηγετικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Βραζιλία δεν θα αναλάβει περιφερειακές πρωτοβουλίες, αλλά δεν επενδύει άμεσα έτσι ώστε να μπορέσει να διαμεσολαβήσει εξ όλων των λατινικών χωρών. Το δεύτερο θέμα είναι καθαρά θεσμικό. Υπάρχουν πολλές ε, επικαλυπτόμενες αρχές οι οποίες είναι φόρα διαλόγου και διάδρασης αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ε, ισχυροί μηχανισμοί για να φτάσουμε σε συλλογικές συμφωνίες. Επίσης, η Λατινική Αμερική δεν θέλει να προσδώσει στα θεσμικά της όργανα το ίδιο ενεργό χαρακτήρα που έχει προσδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικά της. Μας ε, ενδιαφέρει το Μερκοσούρ, η ε, νέα ένωση του ειρηνικού και των χωρών της κεντρικής ε, Αμερικής, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες, δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλους παγκόσμιους φορείς. Αυτό δεν είναι ένα ανυπέρβλητο πρόσκομα για συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφαλείας. Μας ενδιαφέρει η διάδραση μεταξύ Βορείου Ατλαντικού και οργανώσεων της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Επίσης υπάρχει συνεργασία μεταξύ Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενδεχομένως συμμετοχή του ΝΑΤΟ. Η οικονομική συνεργασία θα μπορούσε να προωθηθεί καλύτερα μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτή είναι μεγάλη φορή. Το θέμα δεν είναι δυνατότητα, η δυνατότητα συνεργασίας, αλλά η νομιμότητα. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν αυτές, ε, αυτοί οι μεγάλοι θεσμοί μακροχρόνια. Όμως υπάρχουν προσκόμματα στη διεύρυνση της διατλαντικής συνεργασίας αν δεν επέλθουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει ε, ένα προσχέδιο έτσι ώστε να προωθηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική θέληση για να δεχτούμε την ανάγκη αλλαγής, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το ίδιο θα μπορούσε να αλεχθεί και για τα Ηνωμένα Έθνη Χρειάζεται μεταρρύθμιση και των θεσμών των Ηνωμένων Εθνών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ε, επιρροή ε, και επίδραση στις ε, διατλαντικές σχέσεις. Μέσω των ε, επιμέρους φόρα μιλάμε και για την θαλάσσια ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, την βιωσιμότητα και όλους τους τομείς όπου υπάρχει συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών στο Νότιο Ατλαντικό. Θα πρέπει να χτίσουμε με βάση το διαθέσιμο υλικό. Ζητήθηκε να φτάσουμε σε συστάσεις από την μελέτη μας, όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για άλλους φορείς. Ορίζουμε πέντε στρατηγικά στοιχεία συστάσεων και βεβαίως υπάρχουν και φιλοδοξίες πέρα από το λειτουργικό χαρακτήρα των ε, συστάσεων. Καταρχήν μιλάμε για ενδυνάμωση, ενίσχυση. Εάν η Λατινική Αμερική δεν έχει την ίδια συνοχή όπως η Ευρώπη, ο Καναδάς και η ΕΠΑ, θα πρέπει να αλλάξει αυτό για να υπάρχει ίση εταιρική σχέση θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη Βραζιλία που έχει ηγετική θέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με τη Βραζιλία από το 2007 και υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ε, πολυεθνή και πολυμερή φόρα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ο ηγετικό ρόλος όμως τη ε, Βραζιλίας θα γίνει αποδεκτός αλλού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν οι περιφερειακές οργανώσεις στη Λατινική Αμερική έτσι ώστε να έχουν ενία φωνή. Στην Κίνα και, με την Κίνα και την Ινδία ιδιαίτερα θα πρέπει να προωθήσουμε πολυμερή διάλογο. Η νέα διατλαντική σχέση όμως είναι ένα μέσο και όχι στόχος. Και εδώ μπαίνουν ε, οι άλλες συνιστώσεις. Θεωρούμε ότι μια ευρύτερη διατλαντική σχέση θα πρέπει να αναγνωρίσει τα προβλήματα της περιοχής, να ενισχύσει την διαφάνεια και την ροή πληροφοριών που αποτελεί ε, βασική αρτηρία δραστηριοτήτων και θα πρέπει να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου. Ως προς την ε, βιωσιμότητα θα υπάρχει καλύτερος επιμερισμός άχθους, ιδιαίτερα ως προς τις κλιματικές αλλαγές, την ενέργεια και το περιβάλλον. Θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές με βάση αυτά αποδεικτικά στοιχεία και ε, μία διαδικασία έρευνας και διερεύνησης εκεί όπου χρειάζονται αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να τονίσουμε και τον ε, ανθρώπινο παράγοντα της, ε, μετα, στον τομέα της μετανάστευσης ιδιαίτερα. Θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση, αλλά επισύρουμε την ε, προσοχή και στους ε, φορείς σταθερότητας όπως η ΜΚΟ που μπορούν να λογοδοτήσουν καλύτερα. Η τελευταία συνιστόσα λαμβάνει υπόψη την πρόκληση της συνεργασίας ευρύτερα. Θα πρέπει να ορίσουμε όλους τους επιμέρους φορείς οι οποίοι θα μπορέσουν να επιμεριστούν αυτό το άχθος. Και βεβαίως η κυβέρνηση Ομπάμα το έχει τονίσει αυτό. Θα πρέπει να ακούσουμε τις επιμέρους φωνές της Λατινικής Αμερικής για ε, μεταρρύθμιση και θεωρούμε ότι οι περιφέρειες της Λατινικής Αμερικής διαφέρουν από το συμπαγή ε, χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη, ε, το μεγάλο άξονα της ε, Γαλλογερμανικής Συμμαχίας ε, και ίσως θα έπρεπε να βασιστούμε σε αυτό. Η Ευρώπη και οι ΕΠΑ γνωρίζουν τέτοιες εταιρικές μακρόπνοες σχέσεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία διάδρασης με τις χώρες του Νοτίου Ατλαντικού. Γιατί θεωρούμε ότι μία μακρόπνοη εταιρική σχέση δεν χτίζεται σε μία γενιά και μόνο. Πρόκειται για, ένα ευρύτερο, για μια ευρύτερη κοινωνική διαδικασία η οποία μπορεί να αναπτυχθεί πολυπτύχως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Uh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μιλαμών έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον καθηγητή Jones για τη μελέτη και την παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά την δική μου έκθεση, θα ήθελα να πω ότι έχετε ένα έγγραφο εργασίας που ουσιαστικά συνοψίζει αυτή την έκθεση και διαιρείται σε δύο τμήματα όπως και δική μου έκθεση με βάση την εντολή που έλαβα. Αφενός οι κλασικές θα έλεγα διατλαντικές σχέσεις αφορούν κυρίως τη σχέση μεταξύ Washington και Βρυξελών, δηλαδή είπα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει και μια πιο ευρύτερη προπτική, αυτή που μας ανέπτυξε ο καθηγητής Τζόουν. Συνεχίζω λοιπόν αυτά που ακούσαμε και θα περιοριστώ στο πρώτο τμήμα της έκθεσής μου που αφορά την ευρύτερη, την παγκόσμια προπτική. Αυτή, αυτός ο διατελετικός χώρος έγινε της μόδας τα τελευταία χρόνια. Είχαμε think Tank στο Marshall Fund, ε, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Μαροκινή Κυβέρνηση που σε πρόσφατη πρωτοβουλία ε, μίλησε για μια διατλαντική κοινότητα και, και εγκαινίασε και κάποιες, μια διάσκεψη και δεύτερη ακολούθηση τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον λοιπόν το τελευταίο καιρό για την ευρύτερη αυτή προοπτική. Η βασική ιδέα είναι ότι και οι δύο όχθε του Ατλαντικού, όχι μόνο η βόρεια όχθη αλλά και η νότια, έχουν κοινέ προκλήσει. Οπότε θα πρέπει να τι διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το πιο σκόπιμο και χρήσιμο θα ήταν να το κάνουν ε, με συνεργασία, με κοινή ευθύνη. Και αυτή είναι η ανάλυση που επικρατεί, είναι η κρατούσα γνώμη των τελευταίων χρόνων και των μελετών που διαβάσουμε. Και αυτή ευρύτερη, αυτός ο ευρύτερος διατηλετικός χώρος περιλαμβάνει κάποιες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Βραζιλία, η Νιγηρία, η Νότιος Αφρική, το Μεξικό. Δημιουργεί έντονο ενδιαφέρον λοιπόν και όπως είπε και ο καθηγητής Jones, το γεγονός ότι κάποιες ε, χώρες εκτός του Ατλαντικού όπως η Κίνα, η Ινδία ε, φαίνεται ότι αρχίζουν και κατακτούν κάποιο χώρο και στην Ατλαντική ζώνη και έτσι εντάθηκε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τον παγκόσμιο χαρακτήρα του διατλαντικού χώρου και αυτής της ευρύτερης προοπτικής. Οπότε έχουμε μια ευρύτερη ζώνη που συνδέει Ατλαντικό και Ειρηνικό και γι' αυτό είχαμε πολλές πανεπιστημιακούς κύκλους και φορείς και think tanks που ε, μίλησαν για μια μεταρρύθμιση συνολική του Ατλαντικού χώρου και που δεν θα περιορίζεται μόνο στον Ειρηνικό και στην ΑΚΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προνομιακή σχέση μεταξύ ΕΠΑ και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, ε, του, πρωταγωνιστικού του, τους ρόλου στον διατλαντικό χώρο. Προτάθηκε η ανάγκη για μια πιο συνολική διατλαντική προσέγγιση. Οπότε ποιοι θα είναι οι φορείς ε, αυτής της σχέσης, με ποιους θα έχουμε συνεργασία, ποιοι θα είναι οι συνομιλητέ μα, σε ποιου τομεί και με ποιου μηχανισμού. Τώρα, με ποιου φορεί καταρχήν. Όπω είναι φυσιολογικό με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Ε, περιοχές με στενότατους δεσμούς ε, και με τη ΣΥΠΑ και με, τις, ε, ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιστορικούς δεσμούς και όλο και μεγαλύτερους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς. Ε, γι' αυτό μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν ε, υλοποιήθηκε αυτή η συνεργασία σε πάρα πολλού τομεί. Σε ποιου τομεί θα μπορούσαμε να έχουμε σύγκληση και προστιθέμενη αξία, μα είπε ο κύριο Τζόν, στα θέματα τη ασφάλεια, τη ενέργεια, ε, των λαθρεμπορίων, όπλων, ναρκωτικών, καταπολέμηση κλιματικών αλλαγών, αναπτυξιακή στόχη τη χιλιετία, παγκόσμια διακυβέρνηση το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ε, εκεί υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των βόρειων εταίρων για τα θέματα αυτά. Το θέμα του αφοπλισμού επίσης. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τον κύριο Τζόνς. Υπάρχει ευρύτερη προοπτική και υπάρχει φυσικά και οικονομική διάσταση. Και δεδομένως της πληθώρας των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινοαμερικανικών χωρών, ακόμη και με τον Καναδά που έχουμε σχετικές συμφωνίες. Και επίσης ε, η πληθώρα οικονομικών συμφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες της Λατινικής Αμερικής, ναύτα, συμφωνίες με Κολομβία, Περού, Χιλή, με την Κεντρική Αμερική. Αυτή η νέα ε, συμφωνία που διαφαίνεται και που θα αρχίσουν ως οι διαπραγματεύσεις δημιουργεί ένα πραγματικό τρίγωνο μεταξύ ΕΠΑ, ε, Καναδάς, Μεξικού, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών λατινοαμερικανικών χωρών. Οπότε στο μέλλον θα έχουμε μια τριγωνοποίηση ουσιαστικά αυτών των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Δεν πρόκειται να επεκταθώ στο θέμα αυτό, δεδομένου και του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα περιοριστώ στι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και σε κάποια θέματα που είναι σημαντικά για το μέλλον. Τώρα, με τι μηχανισμού, αυτή είναι η δεύτερη πτυχή. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το διαρευνήσουμε αυτό με τους Αμερικανούς μας εταίρους Βόρειας και Νότιας Αμερικής και Κεντρικής και όπως είπε ο κύριος Τζόνς έχουμε την Ουνασούρ, έχουμε άλλους μηχανισμούς ολοκλήρωσης πιο περιορισμένους γεωγραφικά αλλά ίσως με μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης πρόσφατη συμμαχία του Ειρηνικού, η κοινότητα των Άνδεων, ΣΥΚΑΡΑ και Κεντρικής Αμερικής, Μερκοσούρ, Καρικόμ. Επίσης είναι μια προσπάθεια ολοκλήρωσης ε, των χωρών της Καραϊβικής. Οπότε, με όλες αυτές τις ε, δομές πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο συνεργασίας. Γιατί και εμείς ε, και οι Αμερικανοί, οι Βορειοαμερικανοί, έχουμε τις διασκέψεις κορυφής με τις ΕΛΑΚ, και οι, εμείς με τη ΣΕΛΑ και οι Ηνωμένε Πολιτείε με τις τριετής διασκέψεις κορυφής που έχουμε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θα μπορούσαμε και αυτές τις διασκέψεις κορυφής να τις εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα θα έχουμε σύμπτωση το 2015 για τις α, διασκέψεις κορυφής. Αυτά ως προς τη Λατινική Αμερική. Αλλά υπάρχει και άλλος ακρογωνιαίος λήθος των διατλαντικών σχέσεων με ίσως πιο χαλαρούς δεσμούς σε ό,τι αφορά τις αξίες και τις αρχές, αλλά σημαντικός επίσης εταίρος είναι η Αφρική η δυτική πλευρά της, Ατλαντικής, της Αφρικής, η Ατλαντική όχθη της Αφρικής. Εκεί αναφέρθηκε σε, στην ελευθεροπόρια ναρκωτικών, αλλά την Αμερική, Αφρική, ε, ΗΠΑ, ε, και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι τετρά, τετράγωνες οι σχέσεις γιατί ενώνουν και τις τέσσερις πλευρές του Ατλαντικού. Έχουμε επίσης το λαθρεμπόριο όπλων, την πειρατεία, κλιματικές αλλαγές, παγκόσμια διακυβέρνηση, συνεργασία σε θεσμικά ζητήματα. Όλα αυτά τα θέματα, ε, για όλα αυτά τα θέματα η διατλαντική συνεργασία θα επέφερε μια προστιθεμένη αξία. Επίσης έχουμε και με τις αφρικανικές χώρες ε, την ε, ΣΕΔΕΑΟ, έγινε της μόδας με το Μαλί, έχουμε και θεσμικούς μηχανισμούς για διάλογο και με την Αφρική. Και τέλος, ό,τι αφορά την ευρύτερη αυτή ατλαντική προοπτική. Πρόκειται για ένα για μια ανοιχτή έκθεση ουσιαστικά. Βέβαια, εγώ δεν έχω δυνατότητα να συντάξω έκθεση 60 σελίδων όπως ο καθηγητής Jones. Εμείς έχουμε περιορισμούς στη διάρκεια. Είναι περίπλοκο πάντως το θέμα και θα πρέπει να χαράξουμε τις ε, περαιτέρω γραμμέ μια τέτοια διαδηλαδική συνεργασία. Νομίζω ότι οι βασικοί φορεί επικεντρώνονται στο δικό του θεματολόγιο και σε περιφερειακά ζητήματα και δεν υπάρχει ακόμη μια ε, σφαιρική διατλαντική προσέγγιση και ένα διατλαντικό όραμα. Πιστεύω όμως ότι σταδιακά, προοδευτικά θα πρέπει και αυτό το θέμα να το αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε, παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη, αυτή τη συνείδηση ε, του ανήκειν σε μία ενιαία διατελετική κοινότητα. Αλλά ακόμη ε, έχουμε πόρο από μία τέτοια προσέγγιση. Έχουμε λάβει την έκθεση του κ. Τζόνς, θα τη μελετήσουμε περιστατωμένα και πιστεύω θα εμπλουτίσει τη συζήτηση για την έκθεσή μου. Και το δεύτερο τώρα σκέλος της έκθεσης αφορά τις διμερείς, κλασικές διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πρόκειται να σας κουράσω, έχετε το σχέδιο έκθεσης. Πιστεύω ότι η επανεκλογή του Ομπάμα δίνει ευκαιρία για σύσφυξη των σχέσεων. Είναι σημαντικές αυτές οι διμερείς σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα ποιοτικό άλμα εφόσον ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις που μόλις ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες. Επίσης σημαντική είναι και η συντονισμένη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο, σε θέματα εξωτερικά, εξωτερικής πολιτικής και πιστεύω ότι οι παγκόσμιες αλλαγές ε, θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους δύο αυτούς φορείς για να δράσουν από κοινού αντιμετωπίζοντας τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις και τις κλιματικές αλλαγές και έχουμε και στενή συνεργασία για πολλά θέματα επικαιρότητα. Ε, Συρία, Αφγανιστάν, θέματα Κίνα, Ρωσία, Μαλή, Αραβική Άνοιξη. Είναι απαραίτητο ο συντονισμό μεταξύ των δύο βασικών φορέων τη διατλαντική σχέση, των βόρειων, των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μία ε, διατλαντική ε, συμφωνία και ένας χώρος διαλόγου μεταξύ των βασικών φορέων και να δημιουργηθούν οι βάσεις για ένα στρατηγικό διατλαντικό διάλογο. Κάτι που λείπει αυτή τη στιγμή. Έχω επίγνωση της ανάγκης μιας γνήσιας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι αποτελεσματική ώστε να γίνουμε πραγματικός παγκόσμιος φορέας και τέρος και να μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια βρισκόμαστε σε μια περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας και περικοπών και είπα έχουν, υιοθετούν το δόγμα της ε, αρχηγίας ε, ε, από ένα δεύτερο πλάνο. Επίσης έχουμε και το θέμα του DLD που είναι όργανο διακοινοβουλευτικού διαλόγου, το θέμα του διατλαντικού κοινοβουλευτικού διαλόγου. Και επαναλαμβάνω για να μην σας κουράσω μια και έχετε το σχέδιο έκθεσης και μια και έχω εξαντλήσει και το χρόνο μου, να δώσουμε την προτεραιότητα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον προσκεκλημένο μας τον κύριο Τζόνς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο εισηγητές για την εισαγωγή αυτή που κάναν. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η συζήτηση που θα πρέπει να κάνουμε τον επόμενο καιρό. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι δηλαδικές σχέσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται πάντα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΥΠΑ, ΕΕ, αλλά σε ευρύτερο πλαίσιο για να συμπεριλάβουν και τη Λατινική Αμερική. Ε, θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει σε ό,τι αφορά θέματα διακλαδικών εμπορικών σχέσεων να συμμετέχουμε έντονα όχι μόνο σε ό,τι αφορά τελωνιακές σχέσεις με την παραδοσιακή έννοια δηλαδή, αλλά και το μην ε, δασμολογικών φραγμών, γιατί στρατηγικός πώς είναι σημαντικό το θέμα αυτό από πλευρά δημοσιονομικής πολιτικής και είναι σημαντικό πέρα από την ε, ε, διάσταση της ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση των συμφερόντων από πλευρά ε, των διατελετικών σχέσεων, σύνδεση συμφερόντων και στον οικονομικό τομέα λοιπόν. Για να υπάρχουν κανόνες, να, υπάρχουν, να υπάρχει μια αγορά εργασίας διατλαντική, να υπάρχει μια σχέση μεταξύ βορρά και νότου και με τις είπα, αλλά νομίζω ότι δεδομένη τη ε, ταχύτατα μεταβαλλόμενη κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική η διάσταση τη ε, οικονομική ανάπτυξη και της πολιτική ε, ασφάλειας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό καθίσταται πάρα πολύ σαφές, το παρουσίασαν άλλωστε και οι δύο εισηγητές, Θεωρώ ότι αυτή η τελεωνιακή ένωση δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει μια γενική πολιτική βούληση και πίεση. Αν περιοριστούμε σε θέματα εμπορικής πολιτικής και τα αφήσουμε αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρουμε ότι θα αποτύχουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πίεση πίσω από τη διαδικασία αυτή. Ο συνάδελφος Αλαφράγκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή Jones για την παρουσίαση της έκθεσής του και τον συγητή μας, τον κύριο Μιγιάν για το έγγραφο εργασίας του, που με τη γνωστή του πυγμή ε, και γνώση του θέματος μας κάνει μια εισαγωγή σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας. Και φυσικά σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα, τις προηγούμενες εκθέσεις του κυρίου Μιγιάν. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να υπενθυμίσω ε, τα λόγια του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κυρίου Μπαρόζου στις αρχές του χρόνου, που είπε ότι παρά τις ε, ζωφερές προπτικές που ε, χάραξαν μερικές κασάνδρες για το ευρώ και για την κρίση, είπε ότι τελικά το ευρώ ξεπέρασε την κρίση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απέδειξε ότι είναι σημαντικός παράγοντας ε, στο, στο παγκόσμιο προσκήνιο. 500 εκατομμύρια καταναλωτέ, 300 εκατομμύρια χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα και σημαντικό στι εισαγωγέ και εξαγωγέ αγαθών και υπηρεσιών. Επίση, ο πρώτο ε, δωρητή ε, αναπτυξιακή βοήθεια ε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι ΗΠΑ. Χθε συζητήσαμε με του κυρίου Μαρόπο και Μπαρόζο το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και την αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το μόνο κεφάλαιο που αυξάνεται κατά 30% στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και μάλιστα είμαστε στην προ... ήμουνα στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής ε, στο Σαντιάγο της Χιλής και η συμβολή της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 25% γιατί έχουμε ε, πάνω από 100 εκατομμύρια και εκεί καταναλωτές ε, και μάλιστα είναι τεράστια συμβολή τους και στα Ηνωμένα Έθνη. Ο κύριος Μιγιάννη πολύ σωστά μας υπεθύμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει μια συμφωνία σύνδεσης με το Μεξικό και μια στρατηγική συμφωνία σύνδεσης με εμπορική πτυχή. Έχουμε τέτοιες συμφωνίες με τη Χιλή και το Δεκέμβριο ε, γκριν κυρώσαμε τη Συμφωνία Σύνδεση με την Κεντρική Αμερική και την Συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Δυστυχώ με τη Βραζιλία έχουμε μια στρατηγική σύνδεση, χωρί όμω εμπορική διάσταση. Για προφανεί λόγου δεν ήταν δυνατό μέχρι τώρα να συνάψουμε Συμφωνία Σύνδεση ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μερκοσούρ. Και από αυτή την άποψη περνάμε από μια διμερή ατζέντα, από ένα διμερές θεματολόγιο, σε ένα πιο σφαιρικό θεματολόγιο όπου τα θέματα του διμερούς θεματολογίου δεν είναι τα μοναδικά στην σε διάταξη, αλλά αντιμετωπίζονται και τα μείζωνα παγκόσμια προβλήματα. Καταπολέμηση κλιματικών αλλαγών, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ακούσαμε κάποια στοιχεία τους κατανάλωση ναρκωτικών στη ΣΥΠΑ και στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, με τη συζήτηση που γίνεται για την ομοποίηση της κατανάλωσης και παρά τις κριτικές η κατανάλωση της κοκαίνης έχει μειωθεί δραστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούσαμε και τα προβλήματα με, της μετανάστευσης και άλλα ζητήματα που έχουν μια διάσταση σαφώς παγκόσμια. Στο πλαίσιο αυτό όμως θα πρέπει να πούμε κύριε Πρόεδρε με σαφήνεια ότι έχουμε και κάποια νέα στοιχεία της κατάστασης λόγω της παγκοσμιοποίησης. Γιατί δεν είναι πια η, G8 που διακυβερνά τον κόσμο. Ήμασταν στη, στη Μόσχα και εκεί είδαμε την το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών του G20 με τρει χώρε τη Λατινική Αμερική. Κανένα πριν από λίγα χρόνια δεν φανταζόταν ότι η Κίνα θα επένδυε στη Λατινική Αμερική και θα δάνειζε, είπα, και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα, όπως είπε ένα πολιτικό αναλυτή, ε, ο εξυγχρονισμός δεν προέρχεται από τους ουρανοξύστες του Μανχάταν, αλλά από τους ουρανοξύστες της Κίνας, από το, τους ουρανοξύστες της Σανγκάη. Και ο, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου δεν είναι ο Bill Gates, αλλά ο Κάρλος Σλίμ, ένας ε, Μεξικανός. Οπότε οι παράμετροι της σχέσης έχουν αλλάξει αισθητά. Και η Κίνα με πολύ επιθετικό τρόπο διεισδύει στη Λατινική Αμερική. Είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας, ο δεύτερος εμπορικός εταίρος της Αργεντινής μετά τη Βραζίλια. Και όλοι οι αναλυτές λένε ότι μέχρι το 2015 η Κίνα θα εκτοπίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα γίνει ο πρώτος ε, εμπορικός εταίρος της Λατινικής Αμερικής. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος επενδυτής στη Λατινική Αμερική, δεύτερος οικονομικός εταίρος, πρώτος είναι Μερκοσούρ και Χιλή και η Κίνα ε, μας πλησιάζει και σύντομα θα μας ξεπεράσει στο ρόλο αυτό. Έγινε μια πολύ εύστοχη ανάλυση λοιπόν του προβλήματος και θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποιες ε, συμπληρωματικές σχέσεις μεταξύ της διατλαντικής σχέσης που δεν θα πρέπει να είναι ένα διμερές ε, θέμα πια αλλά τριμερές. Και σε αυτό το τρίγωνο το διατλαντικό έχουμε μια, ένα πιο σαφή επιμερισμό δυνάμεων. Είπαμε γιατί είναι όχι μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου αλλά πέραν τούτου δεν έχουμε ίδια καθήκοντα σε αυτές τις τριμερές ε, σχέσεις. Για παράδειγμα, στην, ε, τα κράτη-μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν στο Τέξας. Ε, μίλησε για την προφορά του Τέξας που έχει ο κ. Τζόνς, αλλά μόνο στο Τέξας οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν περισσότερο από ό,τι επενδύει η Ιαπωνία στις 50 πολιτείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που δείχνει τη σημασία που έχει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην, Πολιτείε Πολιτείες και οι εμπορικές ε, και οικονομικές σχέσεις. Οπότε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια συμπληρωματικότητα μεταξύ της Συμφωνίας ε, Ναύτα που συνδέει είπα Καναδά και Μεξικό και με τι συμφωνίες που έχουμε εμεί με Κολομβία, Περού και άλλους ε, Λατινοαμερικάνους εταίρους, ώστε ο επιμερισμό δυνάμεων μεταξύ του διατλαντικού αυτού να γίνει με πιο ισορροπημένο τρόπο. Και από την άποψη αυτή να μην ξεχνάμε και ένα στοιχείο που επισήμανε και ο καθηγητής Τζόουν. του νέου ε, παράγοντε και την ετερογένεια τη διαδικασία ολοκλήρωση στη Λατινική Αμερική γιατί η ΣΕΛΑΚ αντικατέστησε την ομάδα του Ρίο και είναι μια ομάδα που ε, κυρίως ελέγχεται από τη, τη, Λατινική Αμερική. Έχουμε την Ονασούρ, νέο φορέα ή την νέο φορέα, ή την Συμμαχία του Ειρηνικού, επίσης άλλος νέος περιφερειακός παράγοντας. Οπότε η Λατινική Αμερική δεν έχει πια περιφερειακό ρόλο, αλλά κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση του οικονομικού άξονα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Οπότε όλες οι αναλύσεις που θα κάνουμε στο εξή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το νέο στοιχείο για να κάνουμε μια καλύτερη εξορρόπηση αυτή τη διατλαντική σχέση που, παραλαμβάνω, θα πρέπει να περνάει από τι Ηνωμένε Πολιτείε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική. Σα ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry. Ευχαριστώ Πρόεδρε και λυπάμαι που δεν άκουσα τον συνάδελφο Μίλαν Μον γιατί χρειάστηκε να φύγω για λίγο αλλά άκουσα την εισήγηση του καθηγητή Jones και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή του και είμαι βέβαιη ότι είναι συμπληρωματική προς το έργο του συναδέλφου Μίλαν Μόν. Θα ήθελα να τονίσω πόσο υποστηρίζω την όλη ιδέα της τριγωνικής αν θέλετε συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χωρών της Λατινικής Αμερικής και του Νοτιοατλαντικού και ιδιαίτερα τον ρόλο που θα έπρεπε και θα μπορούσε να διδραματίσει η Βραζιλία σε ό,τι αφορά σε θέματα ασφάλειας αλλά και θέματα γενικότερης ρυθμίσης. Ερωτώ λοιπόν τον, καθηγητά, τον καθηγητή Jones, ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυναμικό που μπορεί να προκύψει από την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΙΠΑ ΕΕ, αλλά και από την πιο διευρυμένη αυτή συνεργασία που συμπεριλαμβάνει χώρες της Λατινικής Αμερικής, όλος η ενδιατέρωση της Βραζιλίας σε ό,τι αφορά τη γενικότερη ρύθμιση, όχι μόνο από οικονομικής άποψης και από εμπορικής άποψης, αλλά και από πλευράς ασφάλειας. Αναφερθήκατε στη σημασία της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ Συμφωνώ, νομίζω, για τη Βραζιλία. Το θέμα της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι θεμελιώδες. Και όχι μόνο για τη Βραζιλία. Θα έπρεπε να είναι θεμελιώδες το ζήτημα για όλους μας. Γιατί προφανώς άπτεται θέμα θεμάτων νομιμότητας των δράσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στην ατζέντα τη ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα ασφαλείας τώρα. Μιλήσατε ποιες ε, είναι οι συνέπειες της διείσδυσης των δυνάμεων της Ανατολικής Ασίας, ιδιαίτερα τη Κίνα στην Αφρική. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι στην παρούσα φάση η ΙΠΑ για εύλογους λόγους και από τεχνολογικής άποψης ε, εγκαταλείπουν μία σημαντική βάση στις Αζόρες. Δεν βλέπουμε όμως να επισέρχεται η Ευρώπη. Αντιθέτως και γίνονται προτάσεις να διεισδύσει η Κίνα με την δύναμη που έχει να τοποθετηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Κανείς δεν απαντάει. Ούτε είπα ΙΠΑ φαίνεται να απαντούν, αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή και η Ευρώπη απαντά. Σχολιάστε λοιπόν αν θέλετε το γεγονός αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναπτύξω λίγο παραπάνω τις συστάσεις σας, τις συστάσεις σας σχετικά με το κοινό αυτό εγχείρημα, το οποίο προαπαιτεί να ακολουθήσουμε τις χρηματοοικονομικές ροές που περιλαμβάνονται στο οργανωμένο έγκλημα και στις τρομοκρατικές δράσεις και που βλέπουμε ότι αναπτύσσονται στην Δυτική ε, Αφρική και στο Νότιο Ατλαντικό. Στη ΣΥΠΑ υπάρχει ήδη σχετική νομοθεσία για το σκοπό αυτό και φυσικά γνωρίζουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΙΠΑ στην εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Δεν υπάρχει όμως κάτι παρόμοιο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια θεωρείτε ότι θα ήταν τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας στους τομείς αυτούς. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Έλς. Να σας ευχαριστήσω για τα θέματα αυτά που θέσατε προς συζήτηση σήμερα το πρωί. Αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση κοιτώντα ε, το 2025 και το 2030, ε, αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει την διατλαντική κοινότητα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των ε, παγκοσμίων αρχών στο διατλαντικό σύστημα, φαίνεται ότι πολλά στοιχεία έχουν αναφερθεί, αλλά τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς, κατά πόσο η εμπορική εταιρική σχέση αυτή, η διατλαντική, θα έπρεπε να συμπεριλάβει και άλλες υπηρεσίες, ε, ψηφιακές υπηρεσίες, ίσως καταστεί σημαντικό τύπο, σημαντικός τύπος ε, παγκόσμιας οικονομίας, στην παγκόσμια οικονομία και έτσι δημιουργήσει νέες βάση για νέες διαστάσεις θέματα όπως η ασφάλεια, μεταξύ του ΝΑΤΟ και ημών θεωρώ ότι θα μπορούσαν να εμπλέξουν και τις ΣΥΠΑ. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε διαδικτική δομή στο μέλλον θα εξαρτάται από μια οικονομική βάση ισχυρή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΕ. Αλλά δύο στοιχεία θεωρώ ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε ό,τι αφορά τις αθλητικές χώρες. Αναφέρθηκε από την, τον υποτεταρμοστή του Μαρόκο το, στο τέλη Νοεμβρίου. Καταρχάς, ότι θα πρέπει να οικονομηθούν ε, δίκτυα ένθεν και ένθεν του αθλητικού. παρά δεν έχω διαβάσει τη σχετική έκθεση. Ε, άκουσα την παρουσίασή σας. Θα πρέπει να αναφερθούν ίσως και οι κεντρικές τράπεζες, να κοιτάξουμε και τι γίνεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. μεταξύ του Εθνικού National Intelligence Council και την Ευρώπη και κοιτώντας τι γίνεται σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες τάσεις, νομίζω ότι καταδεικνύεται ποιο είναι το συλλογικό συμφέρον τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι το εξή. Αυτό που μου λείπει είναι το γενικότερο όραμα, αν θέλετε. Μου κάνει εντύπωση γιατί αντί να κοιτάμε περιφερειακές ομάδες εδώ και εκεί, γιατί κανείς δεν ε, προτείνει ένα ατλαντικό ΑΠΕΚ. Νομίζω ότι γίνεται μια σχετική συνάντηση θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, κάθε δύο χρόνο, μια σχετική ε, συνάντηση για να δώσουμε πιο μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα αυτό, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό δεν θα πετύχουμε τίποτε. Αν όμως κανείς δεν έχει όραμα και κανείς δεν ηγηθεί, ίσως θα μπορούσα να κλείσω με το μήνυμα του Πρόεδρου Μπαρόζο που κάλεσε για τη δημιουργία ενός Ατλαντικού δικτύου γιατί πρόκειται για ένα σύστημα ελεύθερη σκέψη. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια οικονομική συνεργασία όπω αυτή τη Ασία και του Ελληνικού, σε ατλαντικό επίπεδο. Γιατί να μην ξεκινήσουμε λοιπόν από τώρα. Μίστερ Mr. Κύριε Μπουτικόφερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για τις ε, δύο παρουσιάσεις. Ο κύριος Μίαν Μόνα μας έκανε μια, μάλλον έχει πολύ ενδιαφέρον έργο να επιτελέσει. Ταυτόχρονα την ε, περαιτέρω διεύρυνση των διευρυντικών σχέσεων όπως τις γνωρίζουμε και παράλληλα μια προσπάθεια νέου ορισμού των διακλαντικών σχέσεων και θέσης των σχέσεων αυτών σε μια νέα βάση. Θεωρώ ότι το έργο αυτό θα πετύχει μόνο αν και οι δύο πλευρές ε, του παιχνιδιού αυτού αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μην προκύψει αντίφαση μεταξύ των δύο στοιχείων αυτών. Και ο κύριος Έλλης και ο κύριος Μιανμάν είπαν ότι δεν υπάρχει μια ένα συνολικό ατλαντικό όραμα. Αυτό είναι προφανές. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ατλαντικό όραμα χωρίς συνεκτική προσέγγιση για την διατλαντική συνεργασία. Θα πρέπει να επιλέξουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Ένας σημαντικός παράγοντας αυτής της ε, ατλαντικής ε, λεκάνης δεν λεφτεί υπόψη ως σημαντική συνιστόσα, δηλαδή η Αφρική, αν δεν ε, τη θέσουμε στο επίκεντρο την Αφρική, αλλά στην καλύτερη περίπτωση την αναφέρουμε μόνο και μόνο επειδή ενδιαφέρονται για αυτήν οι Κινέζοι, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα διαμορφωθεί αυτό το ατλαντικό όραμα. Ο κύριος Μορ μίλησε για το Global Governance ως σημαντικό θέμα. Συμφωνώ. Αν κοιτάξουμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η παγκόσμια κυβέρνηση στο θέμα των ε, πρώτων υλών καταλήγουμε κατευθείαν στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή της Αφρικής. Αυτή η διατλαντική πτυχή λοιπόν και προοπτική θα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλους τομείς. Δεν πρόκειται να έχει την στρατηγική σημασία που ανέφερε ο James Ellis αν δεν διαμορφωθεί σαν μια πανατλαντική πρωτοβουλία που θα λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες. Αυτό το τρίγωνο που ανέφεραν κάποιοι φίλοι, θεωρώ ότι δεν επαρκεί και είναι παροχημένη, γιατί έχει περάσει ο καιρός που ο Βοράς μπορούσε να επιλέξει ποια συνιστόσα από τον Νότο θέλει να συμπεριλάβει στους παγκόσμιους ηγέτες. Είναι τόσο μεγάλη η δυναμική μεταξύ των χωρών του Νότου, ήδη σήμερα και μεταξύ της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής, που δεν μπορεί να ακολουθηθεί πλέον αυτή η προσέγγιση του τριγώνου. Δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει στρατηγική προσέγγιση και θα πρέπει να προσέξουμε, θεωρώ, σε ό,τι αφορά το Διεθνικό Πολιτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα. Αν αυτό δεν παρεμποδέσει, δεν θέλουμε να παρεμποδίσει τη γενικότερη συνολική προσέγγιση θα πρέπει από την αρχή να συμπεριλάβει και τις χώρες της νότιας, του Νότιου Ατλαντικού. Νομίζω ότι ο κύριος Μπρόκ μίλησε για τις διατραπραγματεύσεις για την εταιρική σχέση, για το εμπόριο και την ε, ανάπτυξη. Θα πρέπει να σκεφτούμε εξ αρχής πώς θα ενταχθούν οι συνιστώσεις αυτές προκειμένου να μην α, παρουσιαστεί ως κάτι αποκλειστικό και κλειστό προς τις χώρες του Νοτιού Ατλαντικού. Υπάρχουν ακόμα τρεις παρεμβάσεις, συνάδελφοι. Ήδη βρίσκεται μεταξύ μας, μαζί μας ο κύριος Κριστιαν Μπέργκερ, ο υπεύθυνος της ΕΙΕΔ για τις σχέσεις με την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα ήθελα να περιοριστείτε στις παρεμβάσεις σας στα δύο λεπτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα που είναι εξίσου ενδιαφέρον. Σιβίτς. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, μακάρι αυτούς τους κανόνες που αναγγείλατε τώρα να τους είχατε επιβάλει από την αρχή της ε, συζήτησης, γιατί περικόπτεται το λόγο μόνο από τους επόμενους ε, μιλητές, ενώ οι προηγούμενοι επέλευσαν μεγαλύτερο χρόνο αγόραυσης Ακούσαμε δύο παρουσιάσεις, την παρουσίαση του δ Τζόνς και την παρουσίαση του εισηγητού μας. Και από τις δύο αυτές ε, παρουσιάσεις προσπαθώ να καταλήξω σε, ε, μια, σε έναν ορισμό που νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την κατάσταση. Πιστεύω ότι οι διατλαντικές σχέσεις αναφέρονται κυρίως ε, στις σχέσεις ε, του, το, της βόρειας όχθης του Ατλαντικού. Μπορούμε βέβαια να διευρύνουμε αυτόν τον ορισμό γιατί αναφέρθηκα ε, και η Κίνα, αναφέρθηκε και η νότια όχθη του Ατλαντικού. Είναι προφανής αυτή η διεύρυνση, αλλά ας μην προσπαθήσουμε ε, μιλώντας για το διατλαντικό διάλογο να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι ουτοπικό νομίζω ευκαιρία του διατλαντικού διαλόγου να επεκτηνόμαστε σε τόσο ευρεία ζητήματα. Νομίζω ότι οι ατλαντικές σχέσει περιορίζονται κυρίως στι ΗΠΑ και οι και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά η λέξη ΝΑΤΟ. Κατά τη γνώμη μου, σε θέματα ασφάλειας είναι σημαντικό να αναφερθούμε σε αυτό το θεσμό που έχει πολύ σημαντική διάσταση και ιστορική αλλά και πρακτική. Επίσης, ε, κάτι που είναι προφανές. Σίγουρα υπάρχει κρίση στις βορειοατλαντικές σχέσεις, στα θέματα που αναφέραμε, γιατί οι ΙΠΑ απομακρύνθηκαν από την Ευρώπη. Οι ε, ε, γύρισαν τις πλάτες ε, στην ε, παλιά σύζυγο, την, ε, την Ευρώπη, γιατί φαίνεται ότι φάνηκαν πιο θελκτικές και τελεστικές σχέσεις με νέους εταίρους, όπως η Κίνα, παρά κάποιες απειλές ασφάλειας που, που αναφέραμε. Επίσης, ακούσαμε από το λόγο του Πρόεδρου Ομπάμα που ζήτησε μια σύσφυξη των διατλαντικών σχέσεων. Θα ήθελα να αναφέρω πέντε τομείς όπου είναι κατεπίγουσα ε, η ανάγκη συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τουλάχιστον ε, σε θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού της ελευθερίας. Ο πρώτος βασικός τομέας είναι η οικολογία, το περιβάλλον. Έχουμε μονίμως πρόβλημα με την εκτέλεση της συμφωνίας που έχουμε συνάψει για να εφαρμόσουμε τη δική μας φιλοπεριβαλλοντική περιβαλλοντική του κόσμου στον κόσμο. Επίσης, ε, το θέμα της ενέργειας. Χρειαζόμαστε μια πιο μακροπρόθεσμη πολιτική για την αξιοποίηση του ρηκτού πλούτου και των φυσικών πόρων. Τρίτος σημαντικός τομέας, το διαδίκτυο. Στα θέματα αυτά, είπα, είναι το τρομερό παιδί, το enfant terrible. Και μάλιστα ε, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων για τα θέματα του διαδικτύου μεταξύ ημών και των ε, Αμερικανών. Ε, βέβαια υπάρχει και το εμπόριο, σημαντικό θέμα, αλλά εκεί θα είναι πιο εύκολο να άρουμε κάποια εμπόδια. Επίσης, μιλήσαμε για την κοινή προσέγγιση ε, σε ορισμένα θέματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω το εξής. Αν και οι δύο εταίροι κινητοποιηθούν προκειμένου να υιοθετήσουμε μια κοινή γραμμή και μια κοινή πολιτική, τουλάχιστον για ορισμένα θέματα όπως τη Μέση Ανατολή, δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε αποτελεσματικές σχέσεις και αποτελεσματική διεύρυνση των σχέσεων προς την Λατινική Αμερική, προς τη Βραζιλία ε, και πιο πέρα ακόμη και προς τον Ειρηνικό και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια μεγάλη εμβέλεια συνεργασίας και όπως τόνισε και ο κύριος Τζόνς, οι παρόντες μηχανισμοί δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ε, του αιώνα μας. Αναφερθήκατε και ε, τις ε, ε, συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, τις μη αναμενόμενες, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει, να αναλάβουμε ευθύνες και για τη διεθνή συνεργασία, όχι ο καθένας να κοιτάει τη χώρα του. Νομίζω όμως ότι το κλειδί για να προχωρήσουμε είναι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Γι' αυτό και το ευρύτερο αυτό όραμα διατλαντικής συνεργασίας θα είχε μεγαλύτερη αξιοπιστία εάν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για ελεύθερο εμπόριο, για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και όπως είπε και ο συνάδελφος Μίλαν Μπον, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για περισσότερες επενδύσεις ως προς την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, αν θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας. Τώρα η πρόταση για τη σύσταση ενός πολιτικού συμβουλίου για τις διατλαντικές σχέσεις νομίζω ότι την πρόταση αυτή θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Και αυτό αφορά και τη συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως είπαν οι συνάδελφοι. Και κάτι άλλο προς τον καθηγητή, τον κύριο Τζόνς. Μιλήσατε για την πειρατεία, για τα ναρκωτικά και ούτω καθεξής, αλλά όχι για την ασφάλεια του κυβέρνοχώρου, κάτι το οποίο είναι ένα μείζον ζήτημα και μας απασχολεί σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και τους διατλαντικούς νομοθέτες. Θεωρείτε ότι τα προβλήματα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου θα πρέπει να μας απασχολούν, να μας απασχολήσουν, να ζητήσουμε από τους εταίρους μας δηλαδή να ακολουθήσουν ε, ελάχιστες προδιαγραφές ε, καλή συμπεριφορά σε σχέση με τη σύμβαση της ε, Βουδαπέστης όπως έχει εξελιχθεί. Ο κύριος Τάνακ, τελευταίος. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας, ενδιαφέρουν, μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρουν πολύ αυτές οι συζητήσεις ε, ευρύτατης εμβέλειας και θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, διατλαντικές σχέσεις και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Λατινική Αμερική. Εγώ είμαι φίλος της Λατινικής Αμερικής. Βεβαίως είναι και η Καραϊβική με την οποία έχουμε μεγάλους δεσμούς και έχουμε και εδάφη και ε, διοικητικά διαμερίσματα εκεί. Μέσα στα πλαίσια της ε, κοινοπολιτείας υπάρχει μια σχετική γεωμετρία η οποία διέπει τις σχέσεις της Βόρειας και της Νοτιοαμερικής, της Ασίας και της Ευρώπης. Ελοχεύει όμως ένας κίνδυνος ε, σε αυτή τη συζήτηση και ο συνάδελφος Κέλλαμ το ανέφερε. Ε, εάν διευρύνουμε τόσο το θέμα, τότε χάνουμε την ουσία. Θα ήθελα να εστιάσουμε την ε, προσοχή μας σε ένα θέμα, δηλαδή τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης-ΥΠΑ, κάτι το οποίο τονίζει και ο Βρετανικός τύπος πρόσφατα. Θα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ένα 30% μόνο θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χώρα μου και προβλέπεται και δημοψήφισμα τα επόμενα χρόνια γι' αυτό. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ έχουν μεγάλη σημασία και νομίζω ότι ε, μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να έχει τη σχέση που έχει με τη Λατινική Αμερική και με τη Βόρεια Αμερική μόνο αν παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ομπάμα και άλλοι πολιτικοί ε, προώθησαν αυτή την ιδέα της ε, παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τζόνς, το βασικό θέμα το οποίο συζητείτε και όπου αποστέλλονται σύμικτα μηνύματα αφορά την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ινδία, ευρωπαϊκή Ένωσης Ινδίας. Σε αυτά τα πλαίσια της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου, εδώ μιλάμε για ναύτα, για ΕΟΧ, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη μετακίνηση ε, ανθρώπων πληθυσμών σε αυτή την περίπτωση και πώς θα ε, άρουμε το πρόβλημα των γεωργικών επιδοτήσεων, διότι ελέγχθη ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εξαιτίας των ε, αγροτικών επιδοτήσεων. Και μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου δεν θα μπορέσει να λύσει το θέμα των γεωργικών επιδοτήσεων. Πώς θα άρουμε αυτό το πρόσκομα. Ο καθηγητής Τζόνς θα μας δώσει απαντήσεις. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να μας απαντήσετε. Μήπως 7. Ας α, το διαπραγματευτούμε. Ήταν συναρπαστική συζήτηση και σας ευχαριστώ θερμά για τη σοβαρότητα με την οποία την αντιμετωπίσετε και λάβατε μέρος αυτή. Εγώ επικεντρώθηκα κυρίως σχέσεις ε, της Ατλαντικού και αυτό λέω στο τελευταίο βιβλίο μου. Εκεί λέω ότι οι οικονομικές σχέσεις και σχέσεις ασφάλειας στο Βόρειο Ατλαντικό ουσιαστικά πρόλαβαν κάποια σχόλια που μίλησαν για την ανάγκη επανένταξη του ΝΑΤΟ στη συζήτηση, δίνοντα στην οικονομία, στι επενδύσει και προώθηση κοινών προδιαγραφών. Και μελετώντας την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, εντοπίσαμε μια σταδιακή ανικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών επιλύει προβλήματα από μόνη τη. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο δεχόμαστε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει οπωσδήποτε να συνάψει κάποιες εταιρικές σχέσεις. Και η πιο ουσιώδης εταιρική σχέση για την κυβέρνηση Ομπάμα και για τις Ηνωμένε Πολιτείε, τουλάχιστον με βάση την Εθνική Στρατηγική του Μαΐου του 2010 και τις επανειλημμένες δηλώσεις ε, των διπλωματικών, ε, η πιο σημαντική σχέση, εταιρική σχέση είναι η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση αυτής της σχέσης αποτελεί σημαντική πρόκληση και αυτήν πραγματευόμαστε στην μελέτη μας για να δούμε πώς μπορεί αυτή η σχέση να αντιμετωπίσει προβλήματα που από μόνες τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείες ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λέει η έκθεση. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε και άλλους φορείς και άλλους παράγοντες που μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στην εξίσωση, ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματική συνεργασία για να ε, εσωτερικεύσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες που έχουν κάνει τις ε, βορειοατλαντικές, διατλαντικές σχέσεις ε, επιτυχής. Το εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες, το εμπόριο σε τις επενδύσεις, ανταλλαγή πληθυσμών, ε, διαπολιτιστικές, διαπροσωπικές σχέσεις και ούτω καθεξής. Και αναζητώντας πιθανούς εταίρους, στραφήκαμε και προς την νότια πλευρά του Ατλαντικού, τη Λατινική Αμερική. Αποδέχομαι την κριτική ότι θα πρέπει και την Αφρική να την φέρουμε σε αυτό το πλαίσιο, και έχω ε, συνεργαστεί πολύ στενά στο παρελθόν με τον Ρωμάνο τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθώντας να βρούμε ένα μηχανισμό για να φέρουμε την Αφρική πιο ε, ενεργά στο προσκήνιο. Και η ολοκλήρωση που λείπει από τη Λατινική Αμερική λείπει ακόμη ε, περισσότερο από την Αφρική. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε αυτή την Ήπειρο για να ε, διερευνήσει περισσότερους μηχανισμούς συλλογικής δράσης. Έτσι θα έχουμε πολύ πιο αποτελεσματική συνεργασία και με την Αφρική. Και το ίδιο ισχύει και για τη Λατινική Αμερική. Η κυρία Γκόμες έθεσε μια πολύ ε, εύστοχη ερώτηση. Είπε, Ας ξεκινήσουμε με αυτό το, ε, την έντονη εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε σε κανονιστικό επίπεδο, σε αριθμιστικό επίπεδο, ώστε να επεκτείνουμε τα πλεονεκτήματα αυτής της υπάρχουσας σχέσης και προς την νότια πλευρά του Ατλαντικού. Και υπάρχουν εδώ ε, τρεις ε, βασικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα τις ε, υγειονομικές και φυτοοικονομικές προδιαγραφές του συστήματος α, της επισητιστικής αλυσίδας, γιατί εκεί υπάρχει σημαντική ε, διαφορά μεταξύ Βορείου και Νοτιού Ατλαντικού. Και θα πρέπει ε, να το λάβουμε υπόψη, γιατί αναφέρθηκε ότι το θέμα αυτό συζητάται και θα πρέπει μέσα σε 18 μήνες να βρεθεί συμφωνία. Αν δεν βρεθεί συμφωνία για αυτά τα, αυτές τις προδιαγραφές, υγειονομικές και φυτοϊγειονομικές, αν δεν μπορούμε να καταλήξουμε στη συμφωνία για να ενταχθούν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής πιο αποτελεσματικά στο ίδιο σύστημα το υγειονομικό και το φυτοϊγειονομικό, τότε θα καταφέρουμε πραγματικά να ε, επιβάλλουμε ένα οικουμενικό πλαίσιο, μια οικουμενική προδιαγραφή στην οποία θα αναγκαστούν και οι Ινδία και η Κίνα να προσχωρήσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε και για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές ε, ε, για το πώς αντιμετωπίζει την οργάνωση του διαδικτύου οι Ηνωμένε Πολιτείε και το πώς αντιλαμβάνονται την ε, προστασία των δεδομένων οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε παρόλα αυτά ότι και το θέμα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για τις χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές και η ανταλλαγή πληροφοριών και για τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες αλλά και σε θέματα μεταναστευτικά θα πρέπει να δρομολογούνται μέσω του διαδικτύου. Αυτή, αυτός είναι ο βασικός διάβλος. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν προδιαγραφές και στάνταρ ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε ε, βασικές πληροφορίες και να τις εξασφαλίζουμε, να τις διασφαλίζουμε, να τις ε, βάζουμε στο απειρόβλητο ε, εξωτερικών επιθέσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν καταφέρουμε να διαφυλάξουμε κάποια κεντρικά σημεία, νευραλικά σημεία του ίντερνετ, νομίζω ότι θα ενισχύσουμε το θέμα της ασφάλειας. Και μπορούμε και με τις χώρες του Νοτιοατλαντικού να επεξεργαστούμε κάποιες κοινέ προδιαγραφές. Έτσι πολύ πιο εύκολα θα ιδιοποιηθούν και αυτές σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Άλλο ζήτημα αφορά τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και επανέρχομαι σε μία παρατήρηση της κυρίας Γκόμες γνωρίζουμε από το Παγκόσμιο Αντιτρομοκρατικό Αγώνα ότι κάποιες δράσεις ασφάλειας ε, μετά την 11η Σεπτεμβρίου ε, μας οδήγησαν το συμπέρασμα ότι οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές είναι το κλειδί για να εξαρθρωθούν κάποια τρομοκρατικά κυκλώματα που είναι και η αχίλιος πτέρνα κάποιων ε, παγκόσμιων ε, κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος, λαθρεμπορίου όπλων, ναρκωτικών και δουλεμπορίου. Θα, πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για να ξέρουμε όλοι τι ζητούμε. Και μάλιστα το θέμα SWIFT μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, και την, το διατηλετικό διάλογο και να αναμίξουμε και τη Λατινική Αμερική αν θέλουμε να επιτύχουμε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και τέλος, είναι απόλυτο σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει αυτό το σχέδιο. Γιατί έχουμε μάθει από την εμπειρία μας ότι δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Θέλουμε μία πιο διευρυμένη σχέση, μία πιο περιεκτική σχέση. Και πιστεύω ότι η Ατλαντική κοινότητα θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της συζήτησης και επίσης να έχουμε ε, με αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, διάλογο που θα είναι ευρύτερο ε, από τα οικονομικά και επενδυτικά θέματα. Θα πρέπει να διευρύνουμε τη συζήτηση και σε θέματα αναπτυξιακά, ασφάλειας, δημοκρατίας, πολιτικής σταθερότητας και πρόθεση της αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που προσπάθησε να προωθήσει ο Ρωμάνο Πρόντι, ενισχύοντα τη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, αλλά και στην Αφρική, με την Αφρικανική Ένωση. Και αυτή είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την προωθήσουμε και παγκοσμίω. Ξεκινώντα με του εταίρου με του οποίου είναι πιο εύκολη η συνεργασία και σίγουρα η Βορειοατλαντική οι εταίροι έχουν ε, ήδη αυτή τη συνεργασία και οι καλύτερε προοπτικέ διαφαίνονται με του εταίρου τη Λατινική Αμερική. Και για τα συμπεράσματα θα δώσω το λόγο εν συντομία στον εισηγητή Μιγιάν Μον. Παρακαλώ χρόνο φίδου, γιατί θα έχουμε και άλλη ευκαιρία για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για τις υποδείξεις που ήταν άκρος ενδιαφέρουσες. Στην ουσία πρόκειται για δύο θέματα. Καταρχήν οι διατλαντικές σχέσεις ε, που θεωρούνται ως μία απτή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ, κάτι το οποίο μας απασχολεί σε καθημερινή βάση και μία πιο μια ευρύτερη ε, διάσταση που αφορά την παγκόσμια προοπτική. Πρόκειται λοιπόν για δύο διαφορετικά θέματα. Ως προς το πρώτο, συμφωνώ ως προς τη σημασία αυτής της έναρξης των διαπραγματεύσεων, ας ελπίσουμε να έχουν αίσιο πέρας και θα ασχοληθώ στην έκθεσή μου με έναν επιμερισμό ε, ευθυνών. Ήδη από τις 3 Οκτωβρίου πέρσι ε, τεθήκαμε υπέρ αυτής της συμφωνίας. Ως προς την ασφάλεια στον ε, κυβερνοχώρο, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2010, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προέβη στη σύσταση μιας ομάδας εργασίας επί του θέματος. Ως προς το Διατλαντικό Πολιτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να το δούμε βαθμιαία θα ήθελα να είχε δημιουργηθεί το 2009 αλλά οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον τότε κρίναν διαφορετικά. Αν θυμάμαι καλά, το 2011 το Διατλαντικό Συμβούλιο ε, μίλησε για διατλαντική ασφάλεια. Δημιουργήθηκε το ΤΕΚ, όπως ξέρετε, το 2007, αλλά δεν διευρύνθηκε η εντολή του. Και η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τάχθηκαν, δεν τάσσονται υπέρ ε, της δημιουργίας νέων φορέων ή οργάνων και ε, εδώ όμως πιστεύω ότι χρειάζεται μία ε, θεσμοθέτηση, μία ειδική θεσμοθέτηση όπως θεωρεί και είπα ύπατη εκπρόσωπος. Θα πρέπει όμως διμερώς να δούμε το θέμα και μετά να ανοίξουμε αυτό το σχήμα σε όλες τις λατινικές χώρες. Θα το δούμε όχι σε αυτή τη θητεία, αλλά σε μία μεταγενέστερη. Ως προς το δεύτερο θέμα, είμαι υπέρ του βαθμιαίου χαρακτήρα. Διότι η, η παγκόσμια θεώρηση του θέματος σημαίνει ότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν ε, βαθμία, διότι οι κυβερνήσεις έχουν άλλες προτεραιότητες και ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική. Τώρα η ΕΠΑ, μάλλον η ΕΠΑ αρχικά, είχαν την προτεραιότητα, είχαν θέσει την προτεραιότητα υπέρ της Ασίας, αλλά νομίζω ότι η διατλαντική προσέγγιση αποτελεί μία από τις δυνατότητες. Αυτό έγινε με το Marshall Fund, το ε, έλαβαν υπόψη και άλλες χώρες. Μιλήσαμε για άλλους σχετισμούς, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και την κόποση, τον παράγοντα κόπωσης των διασκέψεων κορυφής. Απαντώ στον James Ellis. Σήμερα δεν βλέπω ότι οι μεγάλες διασκέψεις μπορούν να αγκαλιάσουν αυτό το θέμα. Βεβαίως, μέσα στα πλαίσια των G20 θα διευρυνθεί το θέμα ή με μια διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν το βλέπω άμεσα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Ο πρόεδρος μου ζητά να είμαι ε, σύντομος και θα το κάνω, όπως σχεδόν πάντα. Σας ευχαριστώ όλους για τις υποδείξεις σας και σας υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα, όλη αυτή η χαρτούρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει και τα όρια της. Σας ευχαριστώ πολύ ως προς το σκέλος της ε, πειθαρχία ε, για τον ε, χρόνο ομιλίας. Ευχαριστώ τον δόκτορα Τζόνς. Περνάμε στο επόμενο θέμα και όπως σας είπα Έχουμε μαζί μας τον Κρίστιαν Μπέργκερ, ο οποίος είναι ε, υπεύθυνος ε, για τις χώρες της Ασίας, του Ειρηνικού, της Αφρικής. Γι' αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε το θέμα της Αιγύπτου και της Τινησίας μέσα στα πλαίσια του Μαγκρέμπ. Όπως ξέρετε στην Αίγυπτο έγινε ένα δημοψήφισμα ενώ στην Τινησία ε, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Μπελαΐντ που ήταν μια σημαντική μορφή της αντιπολίτευσης. Οι χώρες αυτές, ε, η Αίγυπτος και η Τινησία διανύουν μια δύσκολη περίοδο Υπάρχουν ανησυχίε ως προς τη δυνατότητα των ε, κυβερνήσεων να φτάσουν σε δημοκρατικά σχήματα και υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες ως προς τη διακυβέρνηση, θέματα διακυβέρνησης αυτών των χωρών. Μιλάμε για δημοκρατική διακυβέρνηση, η οποία δεν έχει επιτευχθεί και για μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σταματώ λοιπόν εδώ, ζητώντας από τον προσκαλεσμένο μας να μας πει πού βρίσκεται και αν θα λάβει το λόγο. Πού βρίσκεται, α, εκεί. Μπορείτε να παραμείνετε εκεί που βρισκεται εκει μπορειτε να Έχετε το λόγο. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ σήμερα για να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση για την Αίγυπτο και την Τινησία, δύο πολύ σημαντικές χώρες για την συνεργασία. Από ό,τι αναφέρατε και εσείς, ε, οι χώρες αυτές ε, διανύουν δύσκολους καιρούς, ε, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την κατάσταση, όντας όμως σύντομος εισαγωγικά. Θα ήθελα να αρχίσω με την Αίγυπτο, αν μου επιτρέπετε. Βλέπουμε ότι υπάρχει πόλωση πολιτική μεταξύ της αντιπολίτευσης της κοσμικής αντιπολίτευσης και της ε, κυβέρνησης Μόρση. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει δαιμονοποίηση βία στους δρόμους, όπως είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή, για δηλώσεις στο Κάιρο και σε άλλα μέρη στην Αίγυπτο. Και βλέπουμε επίσης ότι, ότι το δικαστικό σύστημα ε, ε, κατηγορείται για τιμωρησία και για αδικίες. Να ξεκινήσω για τα θέματα, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικής μεταρρύθμισης γενικότερα. Είδαμε την ε, διακήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και στα τέλη του προηγούμενου έτους και την επιβολή ε, θραντικών καταδικών μετά τις ε, δίκες, μετά τα περιστατικά στο ποδοσφαιρικό γήπεδο είδαμε έναν νόμο που εφαρμόστηκε για που επιβλήθηκε για την, που επιτρέπει στο στρατό να συλλαμβάνει πολίτες, επίσης την δίωξη δημοσιογράφων, δημοσιογράφων επισήμως για την εξύβριση πολιτικών ατόμων και φαίνεται ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα με τις θρησκείες, με άλλες θρησκείες όπως η Μπαχάη. Είδαμε διαδηλώσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών κατά τις ε, διαδηλώσεις και επιβολής ε, ισχύω ε, και στο Πορτσαΐτ στην διαδηλώσει 27 άτομα έχουν τη ζωή του. Ο κύριος Σταύρος Λαμπρινίτης, ειδικός ε, αντιπροσώπους, μετέβησε στην ε, Αίγυπτο και έκανε καλές συζητήσεις με την ε, κυβέρνηση και ιδιαίτερα με την Προεδρία και επέστρεψε με την εντύπωση ότι υπάρχει βούληση να γίνουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα θέματα που σας ανέφερα και για να Υπάρχει διαβούλευση με τους ε, εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νομοθεσία, ιδιαίτερως για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και για την ελευθερία του συνέρχεσθε. Και πάλι στο τομέα αυτό επιμένουν ιδιαίτερα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και για το δικαίωμα στις, ε, στη διαδήλωση και πάλι αυτό απασχολεί ιδιαίτερα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάτι άλλο θετικό, θετικές ειδήσει είναι ότι η Αίγυπτος έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρατηρήσει τις επερχόμενες εκλογές και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι ότι οι εκλογές θα λάβουν κατά πάσα πιθανότητα χώρα τον Απρίλιο ή αρχές Μαΐου. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία αυτά ακόμα. Σας μίλησα για την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πολιτικό σκέλος, αλλά εξίσου ανησυχητικό, όπως είπατε και εσείς, είναι το σκέλος της οικονομικής διάστασης της κατάστασης, ιδιαίτερα το αυξανόμενο έλλειμμα, η έλλειψη τουρισμού, ο αυξανόμενος αριθμός και ποσοστό, το αυξημένο ποσοστό ένδυα. Τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν πρόσφατα από τον Πεντανίτο Λεώνα, από τον ειδικό αντιπροσώπο τη για τις ε, μεσογειακές χώρε, ο οποίος μετέβησε εκεί την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε συζήτηση βάθο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση για τα θέματα αυτά. Επέστρεψε με ένα σχέδιο για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν κάποια τέτοια θέματα στο μέλλον. Παράλληλα προς τις συζητήσεις αυτές έχουμε και τις συζητήσεις ε, για το δάνειο από πλευρά της Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα από τα πολιτικά κόμματα θεωρεί ότι θα πρέπει να εκδιωχθεί για, για θρησκευτικούς λόγους. Από, πολιτικό, από πολιτική διάσταση τώρα η συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει αναβληθεί με την πεποίθηση ότι χρειάζονται πιο πολλοί συμμετέχοντες σε αυτόν τον εθνικό διάλογο. Θα δούμε τι θα γίνει όμως στο μέλλον. Ένα από τα θέματα τα οποία απασχολεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση είναι κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση εθνικής ενότητας πριν ή μετά τις εκλογές. Η Προεδρία επιμένει ότι η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί μετά τις εκλογές, ενώ η αντιπολίτευση προφανώ θέλει να δημιουργηθεί τέτοια κυβέρνηση εθνικής ενότητας πριν τις εκλογές. Αυτά ως μια πρόγευση των πολιτικών δυσκολιών που, αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, η Προεδρία. Η επίσκεψη των Περνητολαιών ήταν πάρα πολύ σημαντική στο σημείο αυτό, γιατί προσπάθησε να συγκεράσει τις απόψεις αντιπολίτευσης και κυβέρνησης εντόπισε οικονομικούς παράγοντες όπως η ένδια, ο τουρισμός ε, και ούτω καθεξής ως θέματα που απασχολούν εξίσου την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ενδεχομένω να υπάρχει δυνατότητα σύγκληση των απόψεων των δύο πλευρών. Να αναφέρω επίση ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη συνάντηση της Επιτροπής ε, Εταιρικής Σχέσης με την, με την Αιγύπτο εδώ και πολύ καιρό δεν έχει διοργανωθεί σχετική συνάντηση και θέλουμε να καταρτήσουμε και ένα σχετικό σχέδιο για την ε, αποστολή παρατηρήσης των εκλογών. Αυτά σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε αυτά. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους για ερωτήσει. θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι έχουμε ακόμη δύο θέματα το θέμα της ΕΙΕΔ και συμφωνίες εταιρική σχέση και συνεργασίας με κάποιες ε, χώρες της Ασίας. Έχουμε επερπλήρες πρόγραμμα, γι' αυτό θέλω παρακαλώ τους ε, συναδέλφους να περιοριστούν στο 1,5 λεπτό και ε, θέλω να υπολογίζω στην αυρότητά σας. Πρώτα η κυρία Νέιτς. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, Καταρχήν, να θερμά ευχαριστώ στον κύριο Μπέργκερ για τα εισαγωγικά του σχόλια. Μα ζητήσατε να είμαστε λακωνικοί. Θα προσπαθήσω να επισημάνω κάποια θετικά στοιχεία και κάποια πιο ανησυχητικά. Καταρχήν χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι Αιγυπτιακές αρχές έχουν επίσημα προσκαλέσει αποστολή παρατήρηση εκλογών. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από διαφορετικούς προσανατολισμούς και πρίσματα να ενθαρρύνουμε τις επαφές και το διάλογο μεταξύ κόμματος πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης. Και επίσης πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στην Αίγυπτο τη διαλεύκαση κάποιων νομικών ζητημάτων, να δούμε τι περιορισμοί υπάρχουν για τέτοιου είδους παροχή νομικής αρρωγής και αν είναι λογική αυτή οι περιορισμοί. Ελπίζω ο κύριος Λαμπρινίδης να λάβει ενεργό μέρος σε αυτό το διάλογο και να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα, γιατί προς το παρόν Ινστιτούτα και Ιδρύματα και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παρεμποδίζονται στην ε, ε, επιτέλεση του έργου τους. Και επίσης δύσκολη είναι η προσπάθεια και των Αιγυπτιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά έχω κάποιες ερωτήσεις δόθηκε υπόσχεση περισσότερα για περισσότερα. Σε ποιον. Για να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Δεν θα πρέπει να μας απασχολεί μόνο να έχουμε επαφές με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επαφές και να έχουμε στενούς δεσμούς με το λαό της Αιγύπτου πρώτα απ' όλα. Εκεί φοβάμαι ότι κολλησιεργούμε κάπως. Και διαπίστωσα και ανάμεικτα μηνύματα, συγκεχημένα ε, μεταξύ της Λέδη Άστον και του Προέδρου Βαν Ρόμπαϊ. Ποιος είναι ο ρόλος ε, του ενός και του άλλου απέναντι στην Αίγυπτο. Αναφέρθηκε η ετοιμιγορία του Πόρτ Σαΐντ και η καταδίκη σε 21 ατόμων σε θανατική ποινή. Η Λέδη Άστον είπε ότι δεν είπε τίποτα για να καταδικάσει τη θανατική ποινή. Κρίμα που έχασε αυτή την ευκαιρία. Γιατί ανέκαθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της θανατικής ποινής. Γιατί δεν ανέφερε τίποτα η Λέδη Άστον σε μια τόσο σαρωτική ετοιμιγορία και απόφαση. Ε, δυστυχώς παραβιάζονται πλουραλισμός, ε, ελευθερία έκφρασης, ε, χρηστή διαχείριση, κράτος ε, δικαίου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να ενισχύσουμε το ρόλο τους. Αυτό να το επισημάνουμε σε όλες τις επαφές που έχουμε με τους Αιγυπτίους, γιατί αυτά τα θέματα είναι προσφυλέστατα για μας. Και ένα θετικό θέμα. Χαίρομαι που μας προσκάλεσαν για να ε, γίνουμε παρατηρητές σε εκλογές και αυτό ελπίζω να έχει θετικό αντίκτυπο και στη σχετική νομοθεσία για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Χρειαζόμαστε και τα κίνητρα και τα φόβητρα ε, και να είμαστε σαφείς στην οροθετική διαχωριστική γραμμή μεταξύ των κινήτρων και των φοβήτρων, γιατί εκεί υπάρχει μια σύγχυση προς το παρόν. Στις 22 Νοεμβρίου υπευλήθη η πρόταση από 36 βουλευτές ε, της Τινησίας στη συντακτική συνέλευση για τον ποινικό κώδικα. Η πρόταση αυτή των 36 Τινήσεων βουλευτών ε, ε, έχει στόχο την ποινική τιμωρία οποιασδήποτε προσπάθηση εξομάλυση ε, ε, της σιωνιστικής οντότητας εντό εισαγωγικών και να αποφευθεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικών, πολιτιστικών ε, και πολιτικών επαφών με αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως σιωνιστική οντότητα. Και μάλιστα έχουμε και την ε, απειλή φυλάκισης εξαετή και την ε, ε, στέρηση οποιοδήποτε πολιτικού δικαιώματος. Και μάλιστα η πρωτοβουλία αυτή δεν απορρέει από κάποιο μεμονωμένο άνθρωπο, αλλά από μεγάλο αριθμό βουλευτών της συντακτική Συνέλευσης της Τινησίας. Ερωτώ λοιπόν, δεν συνιστά αυτή η πρωτοβουλία μια σοβαρότατη παλινδρόμηση σε σχέση με την πολιτική και την δηλωμένη βούληση της Τινησίας, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι η Τινησία ήταν από τις χώρες του Μαγκρέπ η πιο προηγμένη από την άποψη της δημοκρατίας και της προάσπισης των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη. Κυρία Μπράντον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας κάνατε την ενημέρωση αυτή. Δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Καταρχάς για τον τρόπο που μιλήσατε για την διαδικασία ε, ε, για την σύναψη συμφωνίας ε, εταιρικής σχέσης. Τι θέλουμε να προσφέρουμε και να, για να συνεχίσω από εκεί που τελείωσε η κυρία Σάκε, πού είναι οι κόκκινες γραμμές που θέτουμε, τι θέλουμε να προσθέσουμε και να προσφέρουμε επιπλέον και τι περιμένουμε να λάβουμε σε αντάλλαγμα. Δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά την μαζική ε, καταπάτηση των δικαιωμάτων της, των γυναικών και σε ό,τι αφορά και την αστυνομική μεταρρύθμιση. Σε τι βαθμό βοηθάμε την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά την αστυνομική μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μπέρκερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Το θέμα το θέμα της ε, βοήθειας, της υποβοήθησης για την νομική κατάρτιση. Το συζητήσαμε με τον ειδικό απεσταλμένο για ανθρώπινα δικαιώματα την προηγούμενη εβδομάδα. Μας απέδειξε έντονο ενδιαφέρον η Αιγυπτιακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της ε, εμπειρογνωμοσύνης από ευρωπαϊκής πλευράς και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερω τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την καταγραφή του τι γίνεται και το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά και στο αραβικό πλαίσιο. Και συζητάμε με την, με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση προκειμένου να συνέλθουν και να διαβουλευτούν το συντομότερο δυνατόν οι Ευρωπαίοι υπερογνώμονε με του ε, υπεύθυνου κατάρτιση τη νομοθεσία στο σχέδιο, το τελευταίο σχέδιο τη νομοθεσία για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Τίθεται και πάλι το θέμα της αποδοχής χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές. Αυτό σίγουρα θα μας απασχολήσει τώρα για το more for more που αναφέρατε. Είναι σαφές θεωρώ ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Ε, αναφέραμε πάντα ότι με τα νέα καθεστώτα στην Βόρεια Αφρική συζητάμε, αλλά πάντα διευκρινίζοντας ότι χρειάζεται να διατηρούνται κάποιες αρχές, ο πλουραλισμός, ο πολιτικός και ο σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτά τα θέματα διαρκώς επαναλαμβάνονται και στις συζητήσεις με τις Αιγυπτιακές αρχές αναφερθήκατε ε, και στον Πρόεδρο Φαρόμπα και στην Ελέδη Άστον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επαναλαμβάνουν πάντα τα θέματα αυτά. Μας ρωτήσατε για τον συγκεκριμένο ρόλο των δύο αυτών ε, πολιτικών ηγεσιών. Για την ότι εκπρόσωπο είναι σαφές ότι ηγείται του πολιτικού διαλόγου με την Αίγυπτο και της ε, Task Force, της ομάδας κρούσης με την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων το θέμα της αντικης καταδίκης ε, αναφέρθηκε. Νομίζω ότι πάντα ε, κάνουμε και προβαίνουμε σε δηλώσεις σε περίπτωση επιβολής και εφαρμογής κατα... θανατικής καταδίκης. Και εδώ λοιπόν ε, πολιτικός ε, έχουμε ανταλλάξει απόψεις με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την θανατική καταδίκη. Το θέμα του καρότου, του κίνητρου και του αντικίνητρου είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί στην παρούσα φάση αυτό που προσφέρουμε στην Αιγύπτο είναι η απάλυνση του άχθους ε, των ευάλωτων ομάδων. Συζητάμε ακόμα με την Αίγυπτο θέματα περαιτέρω, όπως για παράδειγμα αυτά που συζητιούνται στα πλαίσια της Επιτροπής Εταιρικής Σχέσης. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κράτους δικαίου και που βρίσκεται η Αίγυπτος. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Σε ό,τι αφορά και τα κονδύλια. Και μπορεί να ενταχθούν στο πλαίσιο της αρχής more for more. Μιλάμε για 90 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το πόσο εξετάζεται. Το ερώτημα τώρα που τέθηκε για τον ποινικό κώδικα της Τινησίας. Από τότε που αναφέρθηκε αυτό στο άρθρο 27 του σχεδίου συντάγματος, το θέσαμε αυτό και στον πρόεδρο της Τινησίας, στον πρόεδρο της σχετικής ε, συνταγματικής επιτροπής της Τινησίας και μας διαβεβαίωσαν ότι το άρθρο αυτό, 27, δεν επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα. Νομίζω ότι η Τινήση ομολογεί. Το ακούν αυτό και από εμάς ως μήνυμα, αλλά και από τη ΣΥΠΑ και από άλλους συνομιλητές και είναι σαφές ότι ένα άρθρο όπως αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό. Για το θέμα της ε, Επιτροπής ε, Εταιρικής Σχέσης, δεν νομίζω. Σύνδεσης. Δεν νομίζω ότι εξέφρασε ικανοποίηση, δεν είναι και πολύ ευτυχή γεγονότα, ξέρετε, οι επιτροπέ αυτέ. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι το εξή, ότι μετά από δύο χρόνια διακοπή των σχέσεων έχουμε μια νέα τέτοια ε, συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να τα θέσουμε τα θέματα αυτά για τους λόγους ακριβώς που αναφέρατε ότι στην Επιτροπή Σύνδεσης θέλουμε να θέσουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Θα πρέπει να ορίσουμε την ε, δομή της Επιτροπής των Υποεπιτροπών που θα εξετάσουν τα θέματα αυτά με σχολαστικό ενδεχομένως τρόπο, αλλά αυτό είναι απαραίτητο για την οικονομική μεταρρύθμιση στην Αίγυπτο. Το θέμα λοιπόν των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σίγουρα θα συμπεριληφθεί στις συζητήσεις, αναφέρθηκε άλλωστε και εδώ. Θα συμπεριληφθεί λοιπόν στη συζήτηση τη επόμενη εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο για τι πληροφορίε που μα ε, δώσατε. Όλο ιδιαίτερο. Θαύμασα το πόσο ε, εκφραστικά μιλάτε τη μητρική σας γλώσσα. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το οποίο και είναι η αναθεώρηση της ε, ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Είναι εδώ ο συνάδελφο Γκουαλχέρι, άραγε, που είναι συνεισηγητή. Να πω δύο λόγια εισαγωγικά. Έχουμε εδώ ένα issue paper. Έχουμε προχωρήσει σε ό,τι αφορά και την κατάρτιση της έκθεσης ε, στη σημερινή συνεδρίαση ωστόσο. Θα θέλαμε εσείς να μας ε, πείτε ποιες παρατηρήσεις θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μετά από την ακρόαση της 28 η Ιανουαρίου. Δύο ακροάσεις έγιναν γιατί θεωρώ ότι και η ακρόαση με τι ε, προξενικέ αρχές αποτελεί τμήμα της όλης διαδικασία. Η αναθεώρηση λοιπόν αυτή της υπηρεσία εξωτερική δράση ε, βρίσκεται σε μία φάση όπου διαπιστώνουμε μεν ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει το εγχείρημα γιατι μία τέτοια ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης χρειάζεται και κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου να καταστεί πλήρως λειτουργική και υφίσταται δύο χρόνια ουσιαστικά και έτσι θα πρέπει πέρα από την κριτική που ασκούμε να είμαστε και δίκαιοι. Τα βέλη της κριτικής έχουν σκοπό να βελτιωθεί η δομή της υπηρεσίας ε, όπως ε, κάνουν άλλωστε προτάσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σκόπιμο λοιπόν είναι να αποφασίσουμε και στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια στη φάση αυτή να διεξάγουμε ένα διάλογο με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο προκειμένου και τα τρία θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στην αναθεώρηση αυτή να προβούν σε μια διαβούλευση. Αυτό ωστόσο θα σήμαινε ότι θα πρέπει να θέσουμε ένα έγγραφο επιτάπητος προς επεξεργασία, προς διαπραγμάτευση. Αυτό αποτελεί μια προσφορά, αν θέλετε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ενδεχομένω στο μέλλον δεν θα προκύψουν αντιφάσεις και συγκρούσεις. Θα το κοιτάξουν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τομείς ε, όπου έχουν ε, καθήλυνα αρμοδιότητα. Η δημοσιονομική αρμοδιότητα τίθεται και θέμα ε, και και θέματα προσωπικού. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση και να υπάρχει και αυτή η ρήτρα αναθεώρησης. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να σας παρουσιάσω αυτή την πρόταση. Η υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης δημιουργήθηκε ως απόρρια, αν θέλετε, της ε, σύμπτυξης τριών ε, υπηρεσιών. Να το έχουμε υπόψη αυτό, της εξωτερικής του Επιτρόπου Εξωτερικών Υποθέσεων, του Υπατορμοστή Σολάνα και του Προέδρου του Υπουργών, του Υπουργού, του Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Αυτές τις τρεις ε, αρμοδιότητες συνενώνει η υπατή εκπρόσωπος. Και διαπιστώνουμε πρέπει να κοιτάξουμε μάλλον κατά πόσον έχουμε πετύχει τις διοικητικές και πολιτικές συνέργειες τις οποίες ε, θέλαμε να πετύχουμε και για τις οποίες δημιουργήθηκε η θέση αυτή. Αυτό αποτελεί για μένα το πιο βασικό. Αυτό αποτελεί τον τίτλο και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε με βάση συγκεκριμένα σημεία. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι υπερβολικά αργές. Και αυτό καθίσταται σαφές και σε ό,τι αφορά την, διαδικασία, ε, εκπαίδευση, την κατάρτιση στο Μαλί. Οκτώβριο αποφασίστηκε αυτό και τέλη Ιανουαρίου διαπιστώσαμε ότι σε τρεις μήνες δεν είχε συμβεί τίποτε. Σε θέματα εφαρμογής δηλαδή. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, τι φταίει. Φταίνε οι δομές λήψεως απόφασης, φταίνε οι ελλείψεις και η αδυναμία επιβολής πίεσης από πλευρά ε, της υπηρεσίας εκδοτική δράσης σε ό,τι αφορά την πίεση, δηλαδή προς τα κράτη-μέλη που έχουν λάβει υποχρεώσεις. Ε, φταίει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση στα κράτη-μέλη, τι φταίει. Νομίζω ότι αυτό εν είδη παραδείγματος καθιστά σαφές ποια είναι τα ερωτήματα. Έχει να κάνει με θέματα διορθωτικής ε, μεταρρύθμισης και πώς μπορούμε να τα αυτοματοποιήσουμε αυτά για να γίνονται πιο γρήγορη τη δικασία. Να δώσουμε κίνητρα. Νομίζω ότι η εμπειρία των τελευταίων μηνών κατέδειξε πόσο σημαντικά είναι τα σημεία αυτά. Τίφεται λοιπόν και ένα θέμα ηγεσία εν γέννη, το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε. Ποια και οι αντιπρόσωποι των εθνικών κρατών μελών είναι σημαντικοί παράγοντες. Αυτό ίσως να καταδεικνύει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές ακόμα. Είμαι βέβαιος ότι ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και πώς δημορφώνεται το προσωπικό του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχει στελεχώσει την υπηρεσία αυτή. Και έτσι τύφεται αυτή η διάσταση, αν θέλετε, μεταξύ διακυβερνητικής και κοινωνικής Ευρώπης. Με ποιο τρόπο μπορούμε, μπορούμε να αποφύγουμε την ε, διοικητική επικάλυψη. προκειμένου η υπατή εκπρόσωπος Μάλλον η υπατή εκπρόσωπος είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Πώς μπορεί έτσι να συμμετάσχει, να συμμετέχει επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ικανοποιητικό τρόπο και Επίσης, αφετέρου, τι γίνεται στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρεί η Επιτροπή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, ως μια ανταγωνιστική υπηρεσία, την οποία ε, δεν θέλει να ενημερώνει για να προασπίζει τα δικά της ε, συμφέροντα ή μπορεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό. Επίσης, ένα πολύ πρακτικό ερώτημα σε ό,τι αφορά τις αντιπροσωπίες. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διάσταση την ψυχολογική. Σε κάποιες αντιπροσωπείες οι υπάλληλοι δεν ε, θεωρούν ότι αποτελούν μία ενότητα ε, ανεπίσημα θεωρούν ότι λογοδοτούν σε διαφορετικό αφεντικό ο καθένας. Και αυτό προκαλεί εντάσεις και επιτόπου. Και δεν επιτρέπει τη δημιουργία καλής συνεργασίας. Αυτό σημαίνει, θεωρώ, ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και θέματα δημοσιονομικής ε, λογοδεσίας. Θεωρώ ότι και εδώ τα πήγαμε καλά σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική ρύθμιση. Θεωρείται ότι μόνο ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας μπορεί να προσυπογράψει όταν είναι έτοιμη η επιταγή, γιατί λέμε ότι είναι η μοναδική δυνατότητα να υπάρχει λογοδοσία ή μήπω τα διοικητικά αυτά θέματα και η υπογραφή διοικητικών εξόδων θα να μπορούν να ανατεθούν σε άλλους. Αυτό τι θα προκαλούσε, θα οδηγούσε σε μια κατάσταση όπου ένας πρέσβης όταν δεν είναι διακοπές δεν θα υπάρχουν, θα γίνονται πληρωμές, γιατί δεν θα μπορεί να υπογράφει. Μιλάμε για μικρά πρακτικά ζητήματα, τα οποία όμως δυσκολύνουν πολύ τη ζωή μας. Και το θέμα των δομών που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Α, μισό λεπτό να μείνω στο θέμα τα προσωπικού. Έχουμε το θέμα της γεωγραφικής και της, ε, της γεωγραφικής ισορροπίας και της ισορροπίας μεταξύ των φύλων. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ένα μόνο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Αποδέχομαι φυσικά ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που δεν ε, είναι οριστική ακόμα. Είμαστε σε φάση προετοιμασίας. Το δέχομαι. Αλλά θεωρώ, πέρα από το ποσοστό που ορίζεται για την συμμετοχή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη εκπροσωπούνται υπερβολικά στις θέσεις των εκπροσώπων. Μπορεί να είναι λαθασμένο αυτό το αίσθημα που έχω, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τα ποσοστά αυτά σε ό,τι αφορά εκπροσώπηση των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να σημαίνουν ότι οι μεν κάνουν την έρευνα και οι δε αποφασίζουν και υπογράφουν. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε τα συνολικά ποσοστά. Θεωρώ ότι είναι μεταβατικό το θέμα αυτό και πολύ που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή που έχουν ε, έλθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζονται στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, βρίσκονται σε μια φάση ευελπισίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να επηρεάσουμε τις δομές αυτές, που είναι σημαντικές και άλλα θέματα. Θέματα εκπροσώπησης, πολιτικής εκπροσώπησης των κοινοβουλίων, του Κοινοβουλίου. το θέμα των εκπροσωπήσεων ad hoc. Είναι τεράστια η επιβάρυνση σωματικά και πραγματικά είναι ανέφικτο να ανταποκριθούν στα καθήκοντα αυτά και αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Και ξέρω ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αγανάκτηση σε ό,τι αφορά και την παρουσία της είπα ε, εκπροσώπου στην Ολομέλεια. Το συζητήσαμε και τον Ιανουάριο Είχαμε συμφωνήσει ότι κάθε δύο μήνες θα έρχεται στην Ολομέλεια. Πάντα υπάρχουν φυσικά πολύ σημαντικές ε, συναντήσεις, αλλά από τη Γερμανία να σας πω ότι ο Πρόεδρος πάντα παρίσταται όταν το ζητάει το Κοινοβούλιο. Τέτοια λοιπόν και πολλά άλλα δικαιώματα του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται και στην Συμφωνία της Μαδρίτης και αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη συμφωνία μας ε, για τη δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε λοιπόν όλα, ότι όλα αυτά τα στοιχεία αυτά που αφορούν και την υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο θα τηρούνται σε ό,τι αφορά όλες τις στρατηγικές αποφάσεις θα πρέπει να α, γίνεται διαβούλευση με την Επιτροπή μας. Προτού ληφθεί η τελική απόφαση. Κάτι τέτοιο δεν έχω δει να συμβαίνει ως τώρα. Ή μήπως με το έχω προσέξει, με έχει διαφύγει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε και φυσικά τύχονται και θέματα που έχουν να κάνουν και με τις δομές ε, ε, άμυνας και ασφάλειας, κατά πόσον όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά πόσον όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα προγραμματίσουμε για να έχουμε περιθώριο ελιγμού με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ε, διαχείριση της ε, στρατιωτικής δράσης και της ε, δράσης σε επίπεδο πολιτικής, πολιτικών ενεργειών. Όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστούν με σωστό τρόπο γιατί στην παρούσα φάση ενδεχομένως να έχουμε δυνατότητα αλλαγή των σημείων αυτών. Δεν ξέρω αν σε 4-5 χρόνια θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε, θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε εξίσου τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την ε, κυρία Άστον, η οποία δείχνει μεγάλη δέσμευση και σαφώς θα έχει και δική της άποψη. Θα παίξουν ρόλο αυτά και στις ευρωεκλογές θα αναφερθούν ως αδυναμίες που θα μας οδηγήσουν ενδεχομένω σε μια κατάσταση όπου δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις και για τις προξενικές αρχές. Μάλιστα, αυτά λοιπόν από μέρους μου. Να παρακαλέσω τον Ρομπέρτο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, παρέμβαση του Έλμαρ Μπρόκ όρισε τα βασικά στοιχεία, οριοθέτησε μάλλον την ε, συνεισφορά μας τη γενικότερη στην ε, αναθεώρηση της δομής και της λειτουργίας της ΕΙΕΔ αναθεώρησης που δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει να προωθηθεί η δυνάμη του άρθρου 13 της απόφασης περί της ΕΙΕΔ. Ένα βασικό σημείο σύγκλησης αφορά την αξιοποίηση των καινοτόμων στοιχείων που εμπεριέχονται στην, ε, στα άρθρα της συνθήκης για τους στόχους της ΕΙΕΔ και για να φτάσουμε σε αυτή τη συνεχτική προσέγγιση η οποία μας απασχολεί συχνά που ε, διέπεται από το πνεύμα της συνθήκης. Και αυτό αντικατοπτρίζεται σε διάφορες πτυχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν και τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση. Ο Μπροκ ε, οριοθέτησε το θέμα, γι' αυτό εγώ θα είμαι πολύ πιο συνεκτικός. Θα σταθώ μόνο στα σημεία που θεωρούμε ε, μίζωνο σημασίας εμείς. Καταρχήν το ρόλο της ύπατης εκπροσώπου. Και εδώ είναι διτό το ζήτημα. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την ύπατη εκπρόσωπο να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά της και ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τον συντονισμό της ΕΙΕΔ. Και θεωρούμε ότι ανταποκρίθηκε μέχρι τούδε ανεπαρκώς σε αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε λοιπόν για ενδεχόμενες λύσεις, δηλαδή να προβλεπόταν και ένας αναπληρωτής γενικός γραμματέας ή εν πάση περιπτώσει να εξεύρουμε λύσεις που θα επιτρέπουν στην ύπατη εκπρόσωπο να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά της που είναι στρατηγική σημασίας ε, μέσα στα πλαίσια μίας εκτενούς προσέγγισης ανταπόκριση στα καθήκοντα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τις νομικές συνέπειες, ε, νομικές νομοθετικές συνέπειες αυτού του εγχείρηματος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την ενότητα αυτού του ρόλου, αλλά να ανταποκριθούμε και καλύτερα και ως ευρωβουλευτές και δεν νομίζω ότι η εκπεριτροπής προεδρία είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν και ε, άλλοι δρόμοι που διανοίγονται δυνάμει του άρθρου 33. Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι η ίδια η διάρθρωση της ΕΙΕΔ. Και νομίζω ότι δύο είναι τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Αυτός ο διτός διοικητικός χαρακτήρας που αντικατοπτρίζεται στο ρόλο του Γενικού Γραμματέα και ενός Chief Operating Officer ενδεχομένως και την Ε, μη πλήρη επίλυση του θέματος της διαχείρισης κρίσεων. Νομίζουμε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει ουσιοδός και η Επιτροπή ΣΕΝΤΕ θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οριοθέτηση αυτού του ζητήματος. Και νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να επιλύσουμε και τον ε, χρηματοοικονομικό χαρακτήρα του εγχειρήματος για να δούμε ποια θα είναι και η θέση του Κοινοβουλίου. Ένα άλλο θέμα αφορά τις αντιπροσωπείες, αυτό είναι σαφέστατο και αυτό που έχει σημασία είναι να μην φτάσουμε σε παράδοξα σχήματα. Δηλαδή, να εγγυηθούμε τον ενιαίο χαρακτήρα, την ενότητα της ε, Ένωσης, αλλά να φτάσουμε σε επιμερισμό ευθυνών. Και αυτό που έχει σημασία είναι και το πολιτικό εγχείρημα, του πολιτικού δηλαδή χαρακτήρα και του προσωπικού των αντιπροσωπιών που δεν εντάσσονται στην ΕΙΕΔ. Πέρα από τις διοικητικές διαδικασίες για τις οποίες ε, μίλησε ο Μπροκ. Ως προς το προσωπικό, στο άρθρο 13 της απόφασης, θεωρείται ότι η πλαισίωση αυτή είναι από τα βασικά στοιχεία του εγχειρήματο θα ήθελα όμως να αποσαφηνίσω ένα στοιχείο. Η διαδικασία αναθεώρησης θα πρέπει να έχει ως στόχο να εντάξει και το άρθρο 6 για το προσωπικό, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να ε, αντιταχθούν ε, στον, κανονισμό προσωπικού, κανονισμό υπηρεσιακής ε, κατάστασης, όπως όρισε και η Επιτροπή Γιούρη. Δεν θα πρέπει να υπάρξει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και έλλειψη νομικής βάσης στις τροποποιήσεις αυτές που θα γίνουν στην ΕΕΔ και αυτό αφορά ιδιαίτερα το staff regulation. και τα θέματα απαρίθμησε ο Μπρόκ. Μιλάμε για την ίση εκπροσώπηση των, δύο φύλων, αλλά και την θεσμική ισορροπία που αφορά τους πάντες, όπως συμφωνήθηκε και στη Μαδρίτη. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα όπως η διαδικασία επιλογής και εδώ χρειάζονται καινοτομίες. Τέλος, το, ως προς το θέμα της ε, λογοδοσίας και της εφαρμογής της Συμφωνίας της Μαδρίτης, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά ανοιχτοί έτσι ώστε να ισχύσει πλήρως το άρθρο 218 και το θέμα της λογοδοσίας που συμφωνήθηκε στη Μαδρίτη. Πριν από την απόφαση περί ΚΕΠΑ και ΕΠΑ. Επίσης θα δούμε πώς θα έχει το debriefing του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν επί του παρόντος. Ευχαριστώ. Ωραία, αρχίζουμε με τη συζήτηση. Κύριε Σαλαφράγκα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Γουαλτιέρη για την παρουσίαση που μας κάνατε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί το Κοινοβούλιο συνέβαλε στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην ανάπτυξη αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Γι' αυτό και θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ μεστή προσέγγιση και να μην υπερβάλλουμε ούτε προς την θετική ούτε προς την αρνητική κατεύθυνση κατά την ανάλυση του έργου της ΑΕΔ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν θαύμα η σύσταση της ΑΕΔ, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι το κατά πόσο η ΑΕΔ όπως δημιουργήθηκε και όπως λειτουργήσε μέχρι τώρα, συνέβαλε στην δημιουργία μιας πιο ορατή ε, συνεκτική και αποτελεσματική εικόνα Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Πολύ άριθμε ήταν οι εμπειρίε μα τον τελευταίο καιρό. Είχαμε την κρίση στη Γεωργία, την Αραβική Άνοιξη, τα προβλήματα στη Λιβύη. Γίναμε μάρτυρες της συμμετοχή συμμετοχής της Παλαιστίνης στην UNESCO, παρακολουθήσαμε τη συζητήση στον ΟΗΕ και Είδαμε και τη σύγκρουση στο Μαλί. Δεν πρόκειται να αντλήσω συμπεράσματα από όλα αυτά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της πολιτικής ευθύνης. Έχω την αίσθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε μόνο να προσπαθήσει να διαφυλάξει τα προνόμια του και τις αρμοδιότητές του, αλλά να συμβάλλει ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και από αυτή την άποψη, όπως είπαν και οι κύριοι Βολτέρη και Μπροκ, να βελτιώσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Νομίζω και δώσαμε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό, ότι χρειαζόμαστε ε, στην, ε, ε στις αξιώσεις μας ε, κάποιες, πολιτικού, κάποιες πολιτικές δομές, ένα είδος ε, πολιτικού συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν στους γενικούς γραμματές κάποιοι πολιτικοί εντεταλμένοι, αλλά και ίσως και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να εξασφαλίσουμε αυτέ τι πληροφορίε και την ενημέρωση που διεκδίκησε στη δική του έκθεση ο κ. Μπροκ. Επίση, αυτό το πολιτικό συμβούλιο θα μπορούσε να επικουρείται από ένα κέντρο στρατηγικού προγραμματισμού υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματέα και με συμμετοχή των άλλων Γενικών Γραμματέων που θα δίνουν προτάσει στο Πολιτικό Συμβούλιο, θα εκτελεί τι αποφάσει και θα εξασφαλίζει την ενότητα των δράσεων και τη συνοχή των δράσεων στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Βέβαια δεν έχω ψευδεστήσεις και αυτά πάτες σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη αυτών των πολιτικών στοιχείων, γιατί γνωρίζουμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως ε, η βασική μου ανησυχία κατά τη στιγμή της αναθεώρησης είναι να μην χαθεί η κοινοτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των δράσεων της ΕΕΔ. Όταν ε, ε, εγκρίθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας, όλοι ε, ελπίσαμε για μια κοινοτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή ήταν η φιλοδοξία μας. Και μετά από μια ε, στάθμιση κατάστασης, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι πριτάνευσε η κοινοτική μέθοδος. Μάλλον επικράτησε περισσότερο η διακυβερνητική μέθοδος. Προσοχή λοιπόν. Θεωρώ ότι η εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι αρμοδιότητε για τα δημοσιονομικά θέματα θα πρέπει να περιοριστούν στο κοινοτικό πλαίσιο. Ο κύριο Γουαλτιέρη μα ρώτησε τι θα γίνει με τι γενικέ διευθύνσει που έχουν και αποχρώσεις ε, που έχουν σχέση και με τη δράση ΕΕΔ. Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ή ανάπτυξη, για παράδειγμα. αυτέ οι γενικέ διευθύνσει που έχουν σαφώς κοινοτικέ αρμοδιότητες θα πρέπει να εμείνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλο το θέμα του συντονισμού αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτά μπορούν να τεθούν στην Αντιπρόεδρο μέσω μιας ειδική ομάδας εργασίας. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι το θέμα, το, του, το θέμα της διοντολογίας των υπαλλήλων Πιστεύω ότι υπάρχει μια αντιδιατολογική συμπεριφορά, για να μην πω ενήθικη. Το επισημάνετε κι εσείς. Και παρόλο που θα πρέπει να το ε, αναλύσουμε πιο διεξοδικά και το διαπιστώνουμε στις συζητήσεις που είχαμε για τις απαλλαγές, υπάρχει υπερβολική ε, εκπροσώπηση κάποιων κρατών μελών στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητες στους υπαλλήλου των θεσμικών οργάνων πραγματικά να συμβάλλουν και να ε, στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Δράσης και να μην γίνουμε μάρτυρες αυτής της ε, αποκαρδίωσης ε, και όχι αντιδεδολογικής συμπεριφοράς α, αποθάρρυνσης που έχει σημειωθεί στους υπαλλήλους. Επίσης, ε, θα πρέπει να τηρήσουμε το συντονισμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να στερήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εξουσίες της. Όταν στην πρώτη έκθεση Μπρόκ είπαμε που θα εντάξουμε την ΕΕΔ, η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε να μείνει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώ δεν έγινε κάτι τέτοιο και βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία αντιστροφής ε, πολύ διαφορετική. Γι' αυτό και η βασική μου ανησυχία ε, στα πλαίσια ε, αυτής της συζήτησης είναι να διασφαλιστούν αμή τι άλλο οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κοινοτικά θέματα. Γιατί αν έχουμε μία επανεθνικοποίηση ή εκτοπισμό του άξονα από την κοινοτική διάσταση στη διακυβέρνηση, ε, για να γίνει κάτι τέτοιο τότε τι χρειαζόμαστε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις για τη λειτουργία της ΑΕΔ. Δεν νομίζω ότι όλα είναι μαύρα και αρνητικά. Πολλές δυσκολίες αντιμετώπιση είπατε εκπρόσωπος και μερικές φορές και αντιστάσεις από, το, από τα μέλη του Συμβουλίου. Αλλά εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να δείξουμε την προσήλωσή μας και δαχθούμε υπέρ της ανάγκης που επισημαίνει και η συνθήκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια εξωτερική πολιτική πιο ορατή, πιο συνεπή, συνεκτική και πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω την γλώσσα μου, αν και δεν το συνηθίζω. Νομίζω ότι καλά θα κάνετε λοιπόν να βάλετε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον συνάδελφο Μπρόκ και τον συνάδελφο Γκουαλχέρη για την ε, εργασία τους και για όλες τις ε, παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που μας απευθύνουν. Όπως φαντάζεστε, στην φάση αυτή υπάρχουν πιο πολλές ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια παρατήρηση η οποία συνάδει με αυτά που είπε και ο πρόεδρος Μπροκ, κοιτώντας πόσο περίπλοκο είναι το, πόσο περίπλοκη η κατάσταση, είναι θαύμα, ένα μικρό θαύμα το γεγονός ότι λειτουργήκαν οι υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Ε, γιατί μάλλον το αντίθετο ήταν το πιο πιθανό. Αυτό είναι θετικό. Αλλά δεν επαρκεί. Τις προηγούμενες εβδομάδες μας προκάλεσαν έκπληξη η έλλειψη των ε, πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στο Σαχέλ και στο Μαλί. Θα πρέπει λεπτομερώς να εξετάσουμε τις αιτίε για την έλλειψη της παρουσίας αυτής και μήπως, να εξετάσουμε, μήπως υπάρχουν ε, προβλήματα της ε, υπηρεσία εκτορικής δράσης και στην θέση της ΥΠΑ της Θεωρώ ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη, αλλά Παρά το γεγονός αυτός, η έλλειψη πρωτοβουλίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη σαφές με οδυνηρό τρόπο μάλιστα ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμα να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι θεωρώ ότι καλά θα κάναμε να εξετάσουμε εις βάθος, ε, για παράδειγμα, την ε, λειτουργία των πολλαπλών αντιπροσωπιών. Το ανέφερε και ο συνάδελφος Μπροκ. Μίλησε για θέματα υποχρή... υποχρέωσης ε, ε, λογοδοσίας και το γεγονός ότι ακόμα και το πιο μικρό κονδύλι θα πρέπει να φέρει υπογραφή του επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε στην Επιτροπή μας ότι δεν μπορούμε να ζητάμε και ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πιο αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων και παράλληλα δυνατότητα ελέγχου έως και της παραμικρής λεπτομέρειας. Εάν θέλουμε να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί, θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάπου μπορεί να προκύψουν σφάλματα και λάθη. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι αρκετά σαφές. Δεν το ξεκαθαρίζουμε και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή στον εαυτό μας. Πώς γίνεται, θέλουμε να έχουμε πλήρη λογοδοσία, αλλά και αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Αυτό δεν είναι απόλυτα συμβατό. Τελευταία παρατηρήση για την πρόταση του συναδέλφου Μπροκ. Η ιδέα να γίνει διαβούλευση με το Συμβούλιο και την ύπατη εκπρόσωπο Άστον και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς αξιολογούν οι ίδιοι την, πώς θεωρούν αυτή την αξιολόγηση της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ενδιαφέρουσα ως ιδέα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε στην πράξη. Να το προσπαθήσουμε όμως τουλάχιστον. Ας κάνουμε μια απλή ε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις εμπειρίες ε, όλων των πλευρών. Συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω απεριόριστα, αλλά αυτό ασφαλώς δεν αποτελεί το στόχο μας. Να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για την εις βάθος ανάλυση και ελπίζω να συνεχίσει η ανάλυση αυτή για να βελτιωθεί τελικά η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Νέιτση, στο μικροφόνο. Α, θεωρώ ότι η πρόταση για συζήτηση με την Λέδη Άστον είναι καλή. Η κυρία Γκόμες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά και τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη για την επισκόπηση που μας δώσατε. Καλωσορίζω τα σχόλια των συναδέλφων. Πιστεύω δε ότι η Lady Άστον θα πρέπει να τις αναγνωρίσουμε το έργο που έκανε για τη δημιουργία της υπηρεσίας και το γενικότερο έργο της. Το γεγονός ότι μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στη λειτουργία της υπηρεσίας εκτορικής δράσης. Αυτό δεν ήταν κάτι το αμεληταίο, ξέρετε, δεδομένου και του θεσμικού πλαισίου που υπήρχε και των ε, προβλημάτων που υπήρχαν και σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό που κατάφερε τώρα σε πολιτικούς όρους που έχουμε φτάσει. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Και διαπιστώνω ότι πολύ συχνά εγώ προσωπικά αναγνωρίζω τη συμβολή της κυβέρνησης Ομπάμα και χαίρομαι που υπάρχει η κυβέρνηση του Ομπάμα παρά τα όσα λάθη και τις ασυνέπειες έχουν σημειωθεί. Βλέπουμε μια πνοή καινοτομία και δημιουργικότητα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και σε ό,τι αφορά τις ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και παγκόσμιων υποθέσεων. Τρεις τομείς θα ήθελα να εντοπίσω, μεταξύ άλλων, στους οποίους θεωρώ ότι η επιρροή των ΗΠΑ είναι πολύ σημαντική και σε ό,τι αφορά τις δικές μας δράσεις, αντιδράσεις και σε ό,τι αφορά την έλλειψη δράσης από εμά, σε ό,τι αφορά την ερμηνευτική διαδικασία, καταρχάς ε, στην Μέση Ανατολή, όπου θεωρώ ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε επιρροή από πλευρά μα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει η Λέδη Άστον, δεν αφιβάλλω καθόλου για το ότι κατανοεί το πόσο σημαντική είναι η σύγκρουση αυτή και πόσο σημαντικές είναι οι προκλήσεις και πόσο μας επηρεάζουν. Φυσικά, δεύτερος τομέας η Αραβική Άνοιξη και ένα κεντρικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα των προσπαθειών μας για την κοινωτική διάσταση των προσπαθειών μας είναι η προσπάθεια α, μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ξέρω ότι υπάρχει αντίσταση από τα μόνιμα μέλη κυρίως του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το θέμα αυτό δεν θα πρέπει να το προωθήσει η Υπηρεσία Εξωτερικής δράση και η δηλαδή Άστον συγκεκριμένα ως υπατή εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος. Αυτό δεν περιλαμβάνεται καν στην ατζέντα, ενώ αποτελεί ένα κρισιμότατο ζήτημα. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος Μπρόκ, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχει μεγαλύτερο ρόλο η ύπατη εκπρόσωπος στον συντονισμό των δράσεων των ε, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και σε ό,τι αφορά την πολιτική σε θέματα ανθρωπιστικά και θέματα διεύρυνσης. Εκεί υπάρχουν όντως προσπάθειες συντονισμού. Αυτό δεν συμβαίνει όμως σε θέματα ανάπτυξης, εμπορίου κτλ. Και αυτό αποτελεί αν θέλετε, κραυγαλαία αντίθεση. Η έλλειψη, για παράδειγμα, τέτοιων ε, συντονιστικών δράσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι θέματα δημοσιονομικά θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα, τον σημαντικότερο ίσως, που θα μας πρόξουν σε μια μεγαλύτερη κοινωνική ενοποίηση. Πρόεδρε, αναφερθήκατε στις προξενικές ε, υπηρεσίες εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στη διπλωματική αντιπροσωπεία, εκπροσώπηση, προκειμένου να υπάρχουν κοινή, κοινά ευρωπαϊκά κτίρια για τις διπλωματικές αρχές και ένας άλλος τομέας στον οποίο θα ήθελα να σημειωθεί πρόοδος είναι ο τομέας ε, της ε, κοινής αστυνομική δράση σε θέματα άμυνα και ασφάλειας. Εδώ δεν βλέπω αρκετά αποτελέσματα και είναι τόσο κρίσιμο ο τομέα αυτός για την ε, αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής μας. Τέλος, να μιλήσω για θέματα ευθύνη λογοδοσία, θέματα τα οποία ανέφερε και ο Κολτιέρη και ο Σαλαφράνκα σε ό,τι αφορά την ε, λογοδοσία τεράστια πρόοδο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στην διαδικασία λήψη αποφάσεων και σε προκτακτική φάση. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο. Ο κύριος Γκουαλτιέρη θα πρέπει να φύγει στις 12 και έχουμε και άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Κοιτάξτε, δεν είναι και τελευταία φορά που θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Σας παρακαλώ, παρουσιάστε τις θέσεις σας λίγο πιο σύντομα. Ιδάλλως θα έχουμε χρονική πίεση και δεν χρειάζεται να αιτιολογείτε κάθε σημείο. Μπορείτε να αναφέρετε απλά το σημείο που σας ενδιαφέρει. Βρισκόμαστε σε φάση συλλογής ε, παρατηρήσεων. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ, κυρία Μπράνερ. Κοιτάξτε, ή θα ισχύει μια γενική, ένας γενικός περιορισμός χρόνους, χρόνου ή όχι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι όταν ε, έρθει η σειρά των πράσινων να μιλάμε λιγότερο. Σχόλιο εκτός μικροφώνου του Προέδρου. Κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρος, η κατάσταση είναι η εξής. Έχουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αυτό το συζητήσουμε ή όχι. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή, ξέρετε. Σας παρακαλώ λοιπόν, προσπαθήστε, προσπαθήστε να ολοκληρώσετε σε δύο λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές για την έκθεσή τους. Νομίζω ότι είναι η σωστή προσέγγιση ε, να έχουμε σε προκαταρκτική φάση της συστάσης μας, ώστε να ασκήσουμε κάποια επιρροή. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά μηνύματα της σημερινής συζήτησης είναι ότι και η ΕΕ θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή την αναθεώρηση και να ασκήσει την αυτοκριτική της. Η αυτοκριτική είναι σημάδι ισχύω και επαγγελματισμού. Δεν είναι καθόλου αδυναμία. Και θα είναι ευκαιρία αυτή για την ΕΕΔ να βελτιώσει τη λειτουργία της. Θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί λοιπόν αυτή την ευκαιρία και εμείς το ίδιο. Σε ό,τι αφορά την συνολική προσέγγιση, μια πιο περιεκτική προσέγγιση. Στο έγγραφο της Μαδρίτης μιλήσαμε για μια κατάλληλη δομή. Δεν την έχουμε όμως ακόμη αυτή τη σωστή κατάλληλη δομή. Δεν υπάρχει. Έχουμε CMPD, CPCC, ξεχωριστές από το υπόλοιπο δεν συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό και πολλές καταστάσεις που επισήμανε οι συνάδελφοι ε, διαπιστώνουν αυτά τα κενά. Επίσης έχουμε την, ε, την ομάδα Μιότσο, αλλά και πάλι δεν υπάρχει συντονισμός, ε, ίσως στη ένταξη στην συνολική δομή της ΑΕΔ. Θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε πώς θα εντάξουμε αυτές τις δομές, ώστε να έχουμε μια περιεκτική προσέγγιση σε καταστάσεις κρίσης και σύγκρουσης. Επίσης, για τα εξωτερικά χρηματο... δημοσιονομικά μέσα. Να τα προσέξουμε και να δούμε τη συνεργασία ΕΙΕΔ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια συγχώνευση των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη συνεργασία και τα εξωτερικά θέματα. Είπαμε ότι και η, και Άστον και ο Πίμπαλξ θα υπογράφει. Αλλά από ό,τι ξέρω, μόνο ο Πίμπαλξ υπογράφει. Η Lady Άστον δεν το κάνει. Παρόλο που θα έχει, έχει τέτοιο δικαίωμα με βάση τι αποφάσει μα. Οπότε να δούμε μήπως ε, η απόφαση που λάβαμε δεν ήταν χρήσιμη και σίγουρα δεν εφαρμόστηκε από ό,τι φαίνεται. Χρειάζεται να θεώρησε επίσης ε, η δομή των, των δομών του Τιμ Σε ό,τι αφορά το θέμα των επιτετραμένων, των πολιτικών επιτετραμένων. Είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιους πολιτικούς επιτετραμένους. Δεν μπορεί η κυρία Άστο να είναι πανταχού παρούσα. Γιατί ούτω ή άλλω η συγχώνευση τριών ιδιωτήτων και τριών υποχρεώσεων σε ένα άτομο είναι ανέφικτη. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Επίσης, χρειαζόμαστε μια αναθεώρηση στις προηγούμενες θέσεις και μια πραγματική ε, γενική γραμματεία, ένα πραγματικό γενικό γραμματέα που θα έχει συνολική ευθύνη και το θέμα επίσης του Συμβουλίου να αναθεωριστεί. Και ο Chief Operating Officer να είναι πραγματικά Operating Officer και να μην ανακατεύεται σε πολιτικά θέματα. Επίσης, θέματα διαχείρισης, ε, πολύ σωστές επικρίσεις έχουν ασκηθεί για το κόστος, αλλά και την χρονοβόρα διαδικασία λήψη αποφάσεων. Επίσης, όπως ε, είπε και ο πρόεδρος, σχεδόν τελείωσα. Σχεδόν. Είναι σχεδόν αδύνατο για την Επιτροπή και το προσωπικό να πηγαίνει σε αντιπροσωπείες. Είναι διπλωμάτες των κρατών μελών αυτοί που πηγαίνουν. Είναι άδικο για τους υπαλλήλους και δημιουργείται ε, πραγματικά μια άδικη κατάσταση, μια κατάσταση πολύ αποκαρδιωτική για τους υπαλλήλους. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί επίσης ε, τα δυνατότητα καλύτερη κατάρτιση ε, για να δούμε τι έχει λειτουργήσει σωστά και τι όχι, σε ό,τι αφορά την ισορροπία των δύο φύλων. Η Λέδη Άστον είχε προ... υποσχεθεί ότι θα αυξήσει την παρουσία των γυναικών στην υπηρεσία, αλλά το σχέδιο που μας υποσχέθηκε δεν το είδαμε ακόμη. Πού είναι λοιπόν αυτή η πρόταση που ανήγγειλε η κυρία Άστον. Αλλά και μεγαλύτερη πολιτική βούληση θα πρέπει να δείξουν τα κράτη-μέλη, όπω είπε η κυρία Νέιτσεν. Δεν μπορεί μία δομή να υποκαθιστά μία πολιτική βούληση. Και φυσικά τα κράτη-μέλη όταν θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα δώσουν και μεγαλύτερε ευθύνε στην ΕΕΔ. Πάντω περιμένουμε συνέχιση των συζητήσεων και εντό του Κοινοβουλίου αλλά και με τη Λέιδη Άστον και το Συμβούλιο για την Επιτροπή. εκτός μικροφώνου στην Επιτροπή ε, εξωτερικής, ε, εξωτερικών υποθέσεων. Μάλλον ο συνάδελφος θα μας δώσει ένα υπόδειγμα πειθαρχίας. Συμμερίζομαι ε, αυτά που είπε η κυρία Μπραντνερ, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανταπόκριση σε μια κατάσταση κρίσης. Νομίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα διάρθρωσης ή πως ίσως υπάρχει πλεονάζουσα διάρθρωση. Θα έπρεπε να συγχωνεύσουμε ενδεχομένως όλα τα σχήματα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην κρίση. Υπάρχει μια διάχυση μέσων, ιδιαίτερα στρατιωτικών μέσων, κάτι το οποίο δεν είναι αποδοτικό. Το ουσιώδες πρόβλημα δεν έγινε στην συγχώνευση αυτών των μέσων, αλλά στην, στο συντονισμό τους. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Μιότζο σε σχέση με την ε, κατανομή αυτών των μέσων. Υπάρχουν όμως μέσα, μέσα στα πλαίσια της ε, ΕΠΑ τα οποία προϋπάρχουν και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε να χτίσουμε μια πυραμίδα η οποία φτάνει στην ύπατη εκπρόσωπο και μόνο σε αυτήν. Αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει μια ε, συνυπευθυνότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ε, μια αλυσίδα συνυπευθυνότητας ή από κοινού ευθύνης και ένας ε, αναπληρωτής γενικός γραμματέας δεν επαρκεί για θέματα ασφάλειας. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η κυρία Άστον μπορεί να ανταποκριθεί σε θέματα ΚΕΠΑ και ΕΠΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα συμβούλιο στο Δουβλίνο για θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά κυρία Άστον δεν μπορεί ποτέ να βρεθεί σε αυτές τις ε, άτυπες συνεδρίσεις. Μπορούμε να μιλάμε για ε, το Μάλι, για θέματα που αφορούν την ατζέντα του 2013 και η κυρία Άστον έχει άλλες εργασίες. Αυτό είναι απογοητευτικό, όπως ισχύει και σε εμά. Δηλαδή, μία φορά το μήνα θα μπορούσε να προσέλθει στο, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Είναι συνεδριάσεις που προβλέπονται έξι μήνες πριν και δεν νομίζω ε, ότι θα μπορούσε, νομίζω μάλλον θα μπορούσε να παρευρίσκεται. Υπάρχει ένα θέμα υπερβολικού συγκεντρωτισμού γιατί μιλάμε για συγχώνευση τριών μέσων και ρόλων. Επίσης, η Αντιπρόεδρος ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη και το θέμα των αποστολών και δυστυχώς για αυτές τις αποστολές, αυτές οι αποστολές δεν την χάνουν ε, επιμελητιακής υποστήριξης. Μιλώ για την Αφρική, ε, στον Νίγηρα ή αλλού και δυστυχώς δεν υπάρχει προγραμματισμός ως προς τη μετάβαση, την αποστολή, την κάλυψη ε, εξόδων ταξιδίου, ξενοδοχεία κλπ. Αυτό προϋπάρχει από την εποχή του Σολάνα και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το επιλύσουμε. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με την εεδ έχουμε αποφανθεί, οι ένορκοι αποφάνθηκαν, αλλά τα κράτη-μέλη κρατούν αμφίσιμη στάση και χρησιμοποιούν αυτή τη στάση ως backup στις διαπραγματεύσεις. Η παρέμβαση στο Μαλί ήταν θέμα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ Κάμερον και Ολάντ. Κατανοώ ότι η ύπατη εκπρόσωπος έχει μεγάλες, ε, ε, αντιμετωπίζει μεγάλες εντάσεις και ε, δεν μπορεί να βρίσκεται παρά με το ένα πόδι στο Κοινοβούλιο και το άλλο στην Κομισιόν ως Αντιπρόεδρος και ύπατη εκπρόσωπος και ασχολείται και με ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν είμαστε υπέρ αναπληρωτών ύπατων εκπροσώπων. Είμαστε κατά αυτής της αρχής. Γιατί μπορεί να υπάρξει διάδραση και με το Κοινοβούλιο για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προς αυτή την ε, κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και όχι να ζητάμε αναπληρωτές ύπα τους εκπροσώπους. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αρχέτυπα τα οποία να ακολουθούμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ποιοι βρίσκονται στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας και να μην βασιστούμε σε πρότυπα τύπου Goldman Sachs. Θα πρέπει να το ξαναδούμε το ζήτημα. Και θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σύνδεσμος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάποιος να έχει διοριστεί. Εγώ είχα προετοιμάσει ένα ταξίδι για την έκθεσή μου για το Σαχέλ και δεν ήξερα με ποιον θα μπορούσα να μιλήσω, ποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει και βασίστηκα στο τέλος στις ε, επαφές μου με την Κομισιόν. Δεν υπήρχε σύνδεσμος από την ΕΙΕΔ. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την προστιθέμενη αξία, γιατί υπάρχουν, δεν υπάρχουν ε, αντιπροσωπείες όπως το Παναμά, Μπαρμπέιντος και ούτω καθεξής. Πρόκειται για ε, ιστορικά, ιστορικές κληρονομιές που θα πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα στα πλαίσια των ε, διπλωματικών σχέσεων και επιτετραμένων. Νομίζω θα μπορούσαμε να προσδώσουμε μία ε, πολύ σχηδή προσέγγιση στην Ε.Ε. και περισσότερο πολύπλευρη. Να, να μιλήσω δύο λόγια, να πω δύο λόγια και να πω ότι τα κράτη-μέλη ουσιαστικά ε, θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την υπηρεσία εκτερικής δράσης. Ε, στην παρούσα φάση, με εξαίρεση τη Γερμανία, τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για την υπηρεσία αυτή. Γιατί τα κράτη-μέλη μειώνουν δραματικά τις δαπάνες στην παρούσα φάση και στην εξωτερική δράση και αποσκοπούν και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό είναι δραματικό για όλη την Ευρώπη, γιατί η οικονομική κρίση αφενός η Ευρώπη καθίσταται σημαντικός παράγοντας, ε, καθίσταται λιγότερο σημαντικός παράγοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο αν ε, γίνεται περικοπή των δαπανών αυτών. Ναι. Και αυτό μειώνει τη σημασία μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι κατά πόσον οι χώρες της Ένωσης, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται όντως ε, για τους ε, να συμπεριλάβουν και να αποσπάσουν τους ε, υπαλλήλους τους στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και ξέρω τη Γερμανία. Γιατί αυτό θα περιορίσει σημαντικά τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παγκόσμιου Προσκήνου. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος yes, thank you. rapporteur for budget. Η συγκήτρια για θέματα προπολογισμού, κυρία Νένσκι. Σας ευχαριστώ. Ε, ο ακρογωνιαίο λήθο τη γνωμοδότησή μου στην Επιτροπή Προπολογισμών στηρίζεται στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ΕΕΔ και αφορά τη, το, τη διαχειριστική χρήση 2011 και αναφέρεται τι συνολικέ διοικητικέ δαπάνε. ε, ε περιλαμβάνουν κάποιο σφάλμα σε ό,τι αφορά τα ε, συστήματα ελέγχου. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στις, στις περιπτώσεις που διε, το ελεκτικό συνέδριο. Αλλά ίσως οι αδυναμίες αυτές οφείλονται στη μεταβατική ε, φάση και την ε, μικρή διάρκεια λειτουργίας μέχρι στιγμής της ΑΕΔ. Πάντω η ΕΕΔ θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως ε, το έργο που έχει γίνει στο δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά και τι βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά τις διοικητικέ δαπάνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μεγάλο τμήμα των διοικητικών δαπανών καταλαμβάνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ μακριά από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προσπίσουμε τα δημοσιονομικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την δημιουργία νομικής βάσης για την ΑΕΔ, εκφράσαμε την ανησυχία μας ζητώντας μία δίκαιη και κατάλληλη γεωγραφική εκπροσώπηση όλων των χωρών μελών και σε όλα τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώσαμε με επιμέλεια τα όσα ακούσαμε. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα υποβάλουμε προτάσεις και θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τις προτάσεις των συναδέλφων. Και με βάση τη σημερινή συζήτηση θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε ένα πρώτο σχέδιο κειμένου, το οποίο και θα σας υποβάλουμε. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε σε πρώιμη φάση διάλογο και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, προκειμένου να ενισχύσουμε την πολιτική ε, ευθύνη μας και την πολιτική αρμοδιότητά μας. Ο Ρομπέρτο έχει το λόγο. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Νομίζω ότι όλοι συνεισέφεραν επαρκώς και όλοι συγκλίνουν σε κοινέ διαπιστώσεις με βάση το δικό μας issue paper νομίζω ότι το πλέον εξέχον στοιχείο αφορά την οντολογική υπόσταση της σχέσης μεταξύ ΕΕΔ και Επιτροπής, όπως είπε και ο κύριος Σαλαφράνκα, και αποτέλεσαν το επίκεντρο των πρωταρχικών μας συζητήσεων το 2010. Και το πρόβλημα έχει ως εξής. Εμείς ε, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια στη Μαδρίτη για να φτάσουμε σε, πιο, σε μια πιο διευρυμένη υπηρεσία από αυτή που ήθελε η Επιτροπή, αλλά πιο κοντινή προς την Επιτροπή από ό,τι επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν ε, ένας αναπόφευκτος συμβιβασμός, δηλαδή ε, πρόκειτο για μια υπηρεσία της Επιτροπής αλλά δεν ε, εντάσσεται στην ε, ΚΕΠΑ. Μιλάμε δηλαδή για τον τετραγωνισμό του κύκλου κατά κάποιο τρόπο. Ε, ευρύες ευρύτερες εξουσίες χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της ολίσθησης προς ένα διακυβερνητικό σχήμα. Το θεωρούμε ως, ένα, ως εφαλτήριο για, την, για μια κοινοτικοποίηση. γνωρίζω πλήρως τα θέματα που θέσατε, αλλά δεν θα πρέπει να δώσουμε μία ε, μάταιη μάχη για να φτάσουμε στο τμήμα 3 του προϋπολογισμού, ούτε να συρρυκνώσουμε την υπηρεσία. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το, την ευρύτητα της υπηρεσίας αυτής χωρίς να αμφισβητήσουμε την ε, κοινοτική μέθοδο. Είπαμε λοιπόν ότι η ύπατη εκπρόσωπος θα πρέπει ουσιοδός να είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής μέσα στα πλαίσια ενός συντονισμού. Αλλά δεν σημαίνει ότι αναλαμβάνει, παίρνει τη σκητάλη η Επιτροπή. Απλώς θέλουμε έτσι να εξασφαλίσουμε μία κοινοτικοποίηση. Αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω, αλλά τα ουσιώδη πολιτικά ζητήματα έχουν ε, επιληθεί. Όσον αφορά την ε, ΚΕΠΑ, ο Ντανζόν έχει δίκιο. Δεν μιλάμε για ενοποίηση, αλλά ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να οδηγήσει σε έναν ε, εξορθολογισμό της δομής. Μιλάμε δηλαδή και για μία διάρθρωση αντιμετώπισης των κρίσεων και θα πρέπει να φτάσουμε σε έναν ορθολογικό μηχανισμό η διάρθρωση. Να λάβουμε υπόψη δηλαδή και τον ε, επιχειρησιακό χαρακτήρα της ΚΕΠΑ μέσα στα πλαίσια των στρατιωτικών ε, διαρθρώσεων, της στρατιωτικής διάρθρωσης, αλλά μην, να μην υπάρχει διαχωρισμός. Να λάβουμε υπόψη και τον γεωγραφικό ιστό. Γιατί η διαχείριση της κρίσης ε, προαπαιτεί μία ε, αποφασιστικότητα θα πρέπει όμως, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, να φτάσουμε σε έναν συντονισμό της διαχείρισης των κρίσεων πέρα από την ΚΕΠΑ. Και αυτό αποτελεί μεγάλη καινοτομία την οποία θα πρέπει να ενθαρρύνουμε. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε στη διαδικασία και κλεισμένων των θυρών. Όποιος λοιπόν δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει θα πρέπει να εγκαταλείψει τώρα την αίθουσα για να πούμε στη διαδικασία του επόμενου θέματος και κλεισμένων των θυρών.